Καλώς ήρθατε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, πρέπει να μιλήσω με τον Λάσε Λέτινεν, γιατί είναι μη παραδεκτές κάποιες τροπολογίες. Έχω μια πολιτική ως πρόεδρος. Ξέρετε ότι εγώ αποφασίζω σχετικά με το αν είναι παραδεκτή ή όχι μια τροπολογία. Ε, άκουσα τις συμβουλές ε, της γραμματείας και αποφάσισα. Αλλά φυσικά πάντοτε θέλω να, πριν λάβω την απόφαση να μιλάω με τον εισηγητή. Γι' αυτό και έπρεπε να μιλήσω με τον Λάσε Λέτινεν. Όπως σας είπα, σήμερα δεν θα την ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση του κυρίου Μπραγκέτο για την κινητικότητα των ασθενών. Γιατί η Επιτροπή ΕΜΒΗ ε, απευθύνθηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για τη συζήτηση σχετικά με τη νομική βάση. Επίσης, ως Πρόεδρος Θα μιλήσω και με τον κύριο Σκυγέ σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις Επιτροπές γιατί υπάρχει μια διάσταση απόψεων και πρέπει να το ρυθμίσουμε. Με, αφού μιλήσω με τον κύριο Μπράγετο τον εισηγητή θα το ρυθμίσω το θέμα. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε, αναβάλουμε την ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Μπραγκέτο. Αρχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Λέτινεν. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες εδώ που δεν θα τις ψηφίσουμε. Η 1, η 35 και η 46. Δεν είναι παραδεκτές αυτές ε, αποφάσεις ε, μετά τις συζητήσεις με τη γραμματεία και τον εισηγητή. Άρα δεν θα τις ψηφίσουμε. Αρχίζουμε. Συμβαστική α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σχολή εκτός μικροφώνου. Ναι, όταν σας ζητήσω να ψηφίσετε ηλεκτρονικά θα ψηφίσετε. Δηλαδή όταν ε, είναι μικρή η διαφορά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ως συνήθως. Καταπίπτει 22, 23 και 24. 25 είναι ταυτόσημοι, ψηφίζουμε για αυτές υπέρ. Κατά. Αποχές. Ιδού λοιπόν ηλεκτρονική εξακρίβωση. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ένας περισσεύει από τους σοσιαλιστές, αλλά ούτως ή δεν πειράζει. 20 προς 22 είναι η έκβαση της ε, ψηφοφορίας. Ε, μια αποχή ε, απορρίπτεται. Απορρίπτονται μάλλον. 27 τώρα είπε. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 27 παρακαλώ. Ένας περισσεύει από τους σοσιαλιστές. Ε, ξαναψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 26 υπέρ 18 κατά. Καμία όχι Εγκρίνεται. 26 καταπίπτει. 28 τώρα υπέρ. Κατά. Α, όχι καταπίπτει. Ωραία. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 35 έχει αποσυρθεί. 36 και 37 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. τη 41 δεν θα την ψηφίσουμε. Μήπως θα έπρεπε, γιατί λέει καλύπτεται από τροπολογία 42. Θα την ψηφίσουμε τελικά. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 δεν είναι παραδεκτή 48 υπέρ Τι είπατε κυρία Στάνερ Αποφάσισαμε το αποκοινούμε τον εισηγητή όσα σας είπα ότι δεν είναι παραδεκτή Μα δεν έχετε καμία αιτιολόγηση γιατί δεν είναι παραδεκτή να σας πω η Επίτροπη δεν μπορούμε να ζητήσουμε μάλλον από την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να εισάγουν ένα νομικό εργαλείο. Δεν είναι η δουλειά της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο μπορεί, αλλά δεν μπορούμε εμείς να ζητήσουμε από την Επιτροπή να το ζητήσει από τα κράτη-μέλη. Εμείς μπορούμε ως Κοινοβούλιο να το ζητήσουμε. Αυτό μου είπε η Γραμματεία. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Διορθώνει ο πρόεδρος. 49 εννοούσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ 54-55 μάλλον λέει ο πρόεδρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55 και 56 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58. Κατά τμήματα η ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, από το Calls on the Commission μέχρι το Inspectorates. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, από το End to Carry Out μέχρι το Inspectorates. Υπέρ για το δεύτερο τμήμα. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 και 62 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 66 καταπίπτει. Η πρώτη τροπολογία υπέρ. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε, λάθος έκανε. η 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίστε για την 3 παρακαλώ. Τώρα περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ. Ξαναψηφίστε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Ναι κύριε Κρέμερ. Ε, σοβαρή παρανόηση υπάρχει εδώ με, κυρίως τη μετάφραση προς τα γερμανικά και στα ολλανδικά. Δεν είναι καλή. Σε, αυτό το, σε αυτή την τροπολογία λέμε ότι ότι δεν καλύπτει πλέον από το ρυθμιστικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Ε, δηλαδή μιλάμε για κλαδικές ε, συμφωνίες, όχι μόνο σε μία βιομηχανία, δηλαδή ε, σε μία επιχείρηση. Έτσι φαίνεται όμως από τη, γερμανική μετάφραση τα αγγλικά σας ενοχλούν. Όχι, τα αγγλικά είναι μια χαρά, λέει ο κύριος Κρέμερ. Εμείς βασόμαστε στην αγγλική εκδοχή. Ψηφίστε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 6 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9, 10 και 11 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η 12 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος ψηφίστε ηλεκτρονικά για την 13 παρακαλώ Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά καμία αποχή εγκρίνεται. Οι 14 και 15 είναι ταυτόσιμες ψηφίστη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 και 21 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Καταπίπτει η 18. Πολύ ωραία. Πάμε στην τελική ψηφοφορία ε, του σχεδίου. Όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Περίσευε eh, eh, ένας από τους ε, σοσιαλιστές. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Παρακαλώ. Έχει την ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 42 ψήφισαν. 28 υπέρ. 14 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Λέτινεν. Då har vi kommit till Yeah. Yeah. Yeah. Motion for resolution, which is this? Yes, which is the final. Oral question and then, okay. Det tre delar, ja. Först och Λοιπόν, πρώτα απ' όλα την νομοθετική πρόταση για τις ε, κατευθυντές γραμμές απασχόλησης. Εδώ δεν υπάρχουν τροπολογίες. Νομοθετική πρόταση δηλαδή ότι δεν προτείνουμε αλλαγή των καταθυντηρίων γραμμών. Παρακαλώ, ψηφίστε. Ηλεκτρονικά εννοείται. Ε, Ψήφισαν όλοι πέρας. 45 ψήφισαν. 42 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Δεν κρίνεται το ψήφισμα. Τώρα η προφορική ερώτηση. Υπάρχει μια τροπολογία όπως βλέπετε. Το we το αντικαθιστούμε με το the community and the member states according to their respective competencies. Η κοινότητα και τα κράτη-μέλη με τις, με τις αρμοδιότητες τους. Έσβησε το μικρόφωνο του Προέδρου και δεν ακούμε. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. συγκρίνεται. Και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ. Ξανά παρακαλώ. Ψηφίστε και πάλι. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν 41 μέλη της Επιτροπής, όλοι υπέρ, καμία αποχή, ωραία, εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο, ξέρετε. Πάμε τώρα στην γνωμοδότηση μετά την προφορική ερώτηση. Ένα λεπτάκι να δω τι έγινε με τη συμβαστική τροπολογία. Λοιπόν, τροπολογία 1 από τον Ούντο Μπούλμαν και τους σοσιαλιστές. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Εδώ έχω μία προφορική τροπολογία. λέει εδώ να, να συμφωνήσει το Συμβούλιο για βραχυπρόθεσμα μέτρα σχετικά με την επενδύσει επενδύσεις για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος. income, αυτό με ενοχλεί, αλλά δεν το αποφασίζει αυτό το Συμβούλιο. Και θέλω να πω και καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και τα κράτη-μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να εξασφαλίσουν επαρκή έσοδα ανάλογα με τις εθνικές πρακτικές. Ναι κύριε Μπουσελ Μάθιος. Επί της αρχής αυτό είχαμε συμφωνήσει, αλλά το ε, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές ε, δεν είναι σωστό. Πρέπει να πούμε τα κράτη-μέλη και κοινωνικοί εταίροι βάσει των εθνικών πρακτικών να εξασφαλίσουν, δηλαδή να μετατοπίσουμε το in accordance to national ε, practice. Με αυτή την αλλαγή μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 2, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική α είπε. κατά αποχές εγκρίθηκε. πίπτη 7. Συμβαστική β είπε. κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει και 8 και ε, ψηφίζουμε για, ηλεκτρονικά τώρα για το σχέδιο γνωμοδότης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίστε, ψηφίστε παρακαλώ. Περισσεύει κάποιος από τους σοσιαλιστές. Ξανά παρακαλώ. Αλλά δεν το έχετε μάθει το μάθημά σας. Αυτός που βγάζει την κάρτα ας την αφήσει έξω μέχρι την επόμενη ψηφοφορία, ο κύριος Μπούσελ Μάθιος. Ε, εμείς θα, α, άμα, θα μας ειδοποιήσετε άμα ε, υπολείπεται ένας από το ΕΛΚ πίσω, όχι μόνο όταν περισσεύει, έτσι δεν είναι πρόεδρο. Λοιπόν, ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι πέρας. Ψ Ψήφισαν 44, 41 υπέρ, ε, κανένας κατά, τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Λόγος ο multilingualism. Yes. You want to say something? Yeah, Rupania Orningsvöga. Merci, Monsieur le Διαδικαστικό από την κυρία το Ευχαριστώ. Ε, να ειδοποιήσω τους συναδέλφους ότι η τροπολογία 2 για τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις γλώσσες, τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά δεν είναι μία τροπολογία πολιτιστικού χαρακτήρα είναι μια τροπολογία που σχετίζεται με τα εργαλεία που μπορεί να έχει κάνει στη διάθεσή του ε, για, τα, για το επάγγελμά του. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος διακόπτει ο πρόεδρος στην κυρία Κασχέτου γιατί δεν είναι διαδικαστικό αυτό, είναι δεν συζητάμε εδώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε συμβαστική α, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ε, καταπίπτει η 1 και ψηφίζουμε την 2 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 3 και ψηφίζουμε την 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 και 18 καταπίπτουν. Συμβαστική D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 και 9 καταπίπτουν, συμβαστική ε υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Οι 7 και 8 καταπίπτουν. Ε, 10, η 10, τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά η 11, η 12, η 13 και η 22. Πάμε στη 14. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 19, 20 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα για το σχέδιο γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 44 ψήφισαν, 43 υπέρ, ένας κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Σόγκορ. Next one is... Okay. Ευχαριστώ, uh, the discharge for the budget Τώρα, απαλλαγή, εγώ είμαι ο συντάκτης γνωμοδότησης. Μία τροπολογία υπάρχει της κυρίας Τάουνερ. Ψηφίστε παρακαλώ. Τροπολογία 1 της κυρίας Τάουνερ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Περισσεύει κάποιος από τους σοσιαλιστές. ψηφίστε παρακαλώ. Όμως είναι ψηφοφορία. it's Μα φαίνεται όταν περισσεύει κάποιος. Πέρας. 44 ψήφισαν όλοι υπέρ. Ε, άρα κανείς κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν η έκθεση της κυρίας Κρετή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν έχουμε τροπολογίες. Ψηφίζουμε κατευθείαν Ηλεκτρονικά για το σχέδιο χρωμοδότησης. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρα. 43 ψήφισαν όλοι υπέρ. Και άρα κανείς κατά καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Κρέτη. Ούτε που τη βλέπω βέβαια την κυρία Κρέτη. ανά την. Και φτάσαμε στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Κοτσιλόβου για την ε, ίση μεταχείριση αντρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή ε, επαγγελματική δραστηριότητα, τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 19, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε την 9-11 ε, ομάδα να τις ψηφίσουμε. Όχι, καλά, 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τις υπόλοιπες τουλάχιστον μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί, δηλαδή 10 και 11 Α, ξέχασα την 8. 8, 8 υπέρ. Για την 8 παραπονιώσασταν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα 10, 11, 12, 13 ομαδών υπέρ. 10, 11, 12 και 13. Όχι, 10, 11, 12 διορθώνω πρώτος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 13 υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και κατά πίπτη 14 15, 16, 17, 1 και 2 ομαδών. Θέλετε? Όχι θα τις ψηφίσουμε με μονομένα. 15 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κατά η 3 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε για το Σχέδιο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ τώρα. Όχι από τους σοσιαλιστές. Ξανά παρακαλώ. είναι και αμφιλεγόμενο. Ε, ε, λοιπόν, πέρας. Σαράντα ψήφισαν όλοι υπέρ. Άρα καμία αποχή, κανένας κατά. Σχαρτήρια κύριε Κοτσιλόβο. Yeah, yeah, yeah, but I have no indication anywhere. No. Okay. Mr. Leider. Μάλιστα κύριε Λέιντε. Πρόεδρε, τρέφω μεγάλο σεβασμό για την συνάδελφο Παναγιωτοπούλου, αλλά έχουμε λάβει 10 στις ε, τροπολογίες εχθές, ε, στις 9 παρατέταρτο. Ε, και οπότε τη είδα σήμερα το πρωί γιατί εγώ είχα φύγει ήδη από το κοινοβούλιο. Μα δεν γίνεται να εργαζόμαστε έτσι, δηλαδή να εξετάσω 10 τροπολογίε μέσα σε ένα τέταρτο σήμερα το πρωί, χωρί να μπορώ να κάνω να μιλήσω με του συναδέλφου, να έχω το χρόνο λίγο να το σκεφτώ, να τι εξετάσω. Ε, μετά τη συζήτηση, αφού ήμασταν στην Επιτροπή χτε ε, όλο το απόγευμα, γιατί τι λάβαμε τόσο αργά. Εγώ ζητώ να μην εξετάσουν αυτέ οι 10 τροπολογίε. Μάλιστα, κύριε Παναγιωτοπούλου. Πρόεδρε, μέχρι τις 7 ήταν η προθεσμία. Πριν τις 7 τις στείλαμε εμείς τις τροπολογίες. Vi kommer att rösta om dem eftersom... Θα τις ψηφίσουμε γιατί έχει δίκιο η κυρία Παναγιωτοπούλου. Ναι, η προθεσμία ήταν, ε, ήταν σε 7. Αλλά ε, όπως σωστά είπε ο κύριος Λέιντε δεν είναι ικανοποιητική αυτή η διαδικασία, δηλαδή οι τροπολογίες που δεν έχουν συζητηθεί να τη, καλούμαστε να τις ψηφίσουμε γιατί δεν τις είχαμε ψηφίσει τις τροπολογίες. Επ' αυτό έχει δίκιο ο κύριος Λίντε. Εφόσον όμως υπήρχε προθεσμία, θα τη τηρήσουμε, δεν μπορώ παρά να τις ε, υποβάλω σε ψηφοφορία τις τροπολογίες. Για το μέλλον όμως, κυρίως για τις προφορικές τροπολογίες, ας προσπαθήσουμε να συζητούμε τις τροπολογίες όλες. Δεν ξέρω πώς θα τοποθετηθούν οι πολιτικές ομάδες. Μπορεί Πλώς κάποιο να καταψηφίσει κάποιε τροπολογίες επειδή δεν πρόλαβε να τις διαβάσει και να τι εξετάσει. Έτσι. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Λοιπόν, προφορική τροπολογία. Εν, ε, προφορική ερώτηση τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Μπερδεύτηκα. Ψηφίστε ξανά για την ε, τροπολογία 2. Ξαναλένε η προφορική ερώτηση. Μιλάμε για την προφορική ερώτηση. Τροπολογία 2 για την προφορική ερώτηση. Δεν έχουν αποφασίσει οι πολιτικές ομάδες ε, ε τι θα ψηφίσουν. Ε, συγγνώμη, έχουμε δύο προφορικές ερωτήσεις. Μία προς το Συμβούλιο και μία προς την Επιτροπή. Ε, ποια εννοείται. Προς την... Ε, α, προς την Επιτροπή εννοείται, εντάξει. Γιατί έχουμε... τις έχουμε βάλει με διαφορετική σειρά. Προς την Επιτροπή, τροπολογία 2. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ για την ε, προφορική ερώτηση προς την ε, Επιτροπή. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι πέρας. 41 ψήφισαν, 40 υπέρ, κανείς ε, κατά, μία αποχή εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην άλλη προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, ψηφίζουμε τώρα για την ε, προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Παρακαλώ, ψηφίστε. Άρχιτε ψηφοφορία. Υπέρ. Ε, συγγνώμη, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, 40 ψήφισαν, 38 υπέρ, κανείς κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται επίσης και πάμε τώρα στη γνωμοδότηση. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Όχι λάθος. Για... Δύο. Ναι, εντάξει, λάθος έκανα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 39 ψήφισαν, 17 ε, υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 τώρα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι πέρας 41 ψήφισαν 40 υπέρ Καμία ψήφος κατά, μία αποχή εγκρίνεται. Εντάξει, δεν θα ε, ε, συγχαρώ τον υποφαινόμενο. Ναι, Φίλιπ. Πρόεδρε, ε, ένα διαδικαστικό για την καθυστερημένη υποβολή τροπολογιών Είπατε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Τι δίδαγμα πρέπει να αντλήσουμε από αυτό. Καλό είναι χρήσιμο να συζητούνται οι τροπολογίε στην Επιτροπή, αλλά επίση η Γραμματεία καλό είναι να μα δίνει περισσότερο χρόνο για να υποβάλουμε τροπολογίε. αλλά ένα από τα διδάγματα είναι ότι δεν πρέπει την προηγουμένη στι 7 να είναι η προθεσμία. Εντάξει, να έχουμε ίσω λίγο λιγότερο χρόνο, Δυστυχώ για τι τροπολογίε στο μέλλον. Δίκιο έχετε. Είπα ότι συμφωνώ με τον κύριο Λέιντε γιατί για ε, οποιαδήποτε γνωμοδότηση πολύ καλό είναι να έχουμε συζητήσει τις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε την επομένη. Αυτό είπα. Το θέμα είναι πώς θα ορίσουμε την προθεσμία. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά το σημαντικό είναι να τη συζητούμε τις τροπολογίες πριν τις ψηφίσουμε. Λοιπόν, πέρα των ψηφοφοριών ε, και ε, προχωράμε. Το επόμενο λοιπόν σημείο επέκταση των τύπων δαπανών που είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΚΤ τροποποίηση του κανονισμού 1081 το 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η κυρία Καρίν Γιόνς είναι η συγγήτριά μας ε, και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ στην πρόταση αυτή μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο είναι τμήμα του πακέτου ανάκαμψης και συγκεκριμένα μιλάμε για την ε, διευκόλυνση της ροής των κεφαλαίων ε, του ΕΚΤ και την επιτάχυνσή τους, κάτι το οποίο βεβαίως τώρα απαιτείται κατεπηγόντως. Θεωρώ ότι είναι καλή η πρόταση της ε, Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο εμείς ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή ζητούσαμε πάντα από την Κομισιόν και το Συμβούλιο και βεβαίως είναι λίγο κρίμα πως ε, ειδικά τώρα στην κρίση κάνουν κάτι τέτοιο και λένε εντάξει είμαστε διατεθειμένοι να κινηθούμε λιγότερο γραφειοκρατικά. Να σας πω λίγο περί τίνος πρόκειται. Αυτή τη στιγμή τα εγκεκριμένα μέσα προκαταβάλλονται σε πολύ μικρό ποσοστό και ο νέος ε, κανονισμός αυτός διευρύνει την δυνατότητα καταβολής προκαταβολών στα έργα και να δίνεται μια πληρωμή συνολική κατά για άμεσα και έμεσα έξοδα και να έχουμε κατά αποκοπήν ποσά μέχρι και 50.000 ευρώ που μπορούν να καταβληθούν. Και θα σας το πω ανοιχτά. Ε, δεν ήμουν τόσο σίγουρη στην αρχή, ερχόμενη εγώ από τον προϋπολογισμό, γιατί λέω πρέπει να μπορούμε και να τα ελέγχουμε αυτά. Μίλησα όμως με πολλές εθνικές υπηρεσίες στα κράτη-μέλη και με τους ελεγκτές εδώ του προϋπολογισμού και με την Κομισιόν και πίστηκα πόσο έλεγχος ε, επί της αρχής υπάρχει, είναι δεδομένος το πρόβλημά μου ήταν πως ε, δεν υπήρχε ανώτατο όριο στις πληρωμές αυτές κατά αποκοπήν. Παρόλα αυτά μπορούμε να υπερψηφίσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα γιατί τα κατά αποκοπήν αυτά ποσά και πληρωμές πρώτα απ' όλα θα οριστούν από τα ίδια τα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή μιλάμε για ποσά και ποσοστά που θα ορίσουν τα κράτη-μέλη και πρέπει τον υπολογισμό που θα κάνουν να, να τον υποβάλουν εκ των προτέρων στην Κομισιόν για να τον ελέγξει και αναφέρεται εδώ πως η πρόταση που θα υποβληθεί πρέπει να είναι δίκαιη, ισορροπημένη και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να επαληθευτεί δηλαδή θα τη τηρήσουν και τα κράτη-μέλη και θα υπάρχει πάντα η, ο πρώτος έλεγχος κομισιών και αν ε, βεβαίως δεν συμφωνήσουμε δεν θα προχωρήσουμε χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα τώρα γι' αυτό δεν έχω δεχτεί ε, τροπολογίες και ελπίζω να σας έπεισα και να σας έπεισα να μην υποβάλλετε και εσείς τροπολογίες για να τελειώνουμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, ε, το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα στους συντονιστές. Ε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να προδικάζουμε. Ναι, εντάξει, πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι για την χρήση των κονδυλίων με ικανοποιητικό τρόπο. Ορισμένε φορές χρειαζόμαστε πολύ γρήγορα αυτά τα κονδύλια. Οπότε δεν πρέπει να φαίνεται ότι εμείς το κοινοβούλιο, ότι εμείς από το κοινοβούλιο καθυστερούμε τη διαδικασία. Δεν, ε, δεν πρέπει να δίνουμε αυτή την εντύπωση. Αυτά λέγαμε με τους συντονιστές. Και κάποιοι συντονιστές συμφώνησαν. Αλλά βέβαια, όπως είπε και η κυρία Γιάννησε, θα πρέπει να ε, έχουμε την δυνατότητα ελέγχου. Αλλά τα κράτη-μέλη χρειάζονται, δεδομένης της ε, δυσχερούς κατάστασης, γρήγορα αυτούς τους οικονομικούς ε, πόρους. Η κυρία Στάουνερ τώρα και ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγήτρια κατά βάση. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε εδώ πέρα η κυρία Κύριε Γιάννης, πράγματι πρέπει να βρούμε μια ισορροπημένη λύση. Έχουμε όλη την κοινή πρόθεση, δηλαδή την αποτελεσματική ροή των κεφαλαίων του ΕΚΤ, αλλά απ' την άλλη να υπάρχει και ένας λογικός έλεγχος που δεν θα χρησιμοποιεί όλους τους μηχανισμούς που υπάρχουν να βρούμε μια ισορροπία. Οπότε και εγώ θεωρώ πως χρειαζόμαστε αυτά τα ποσά κατά αποκοπήν γιατί είναι λογικότερο όπως λέω πάντα να μην χρειάζεται να υποβάλουμε κάθε εισιτήριο του τραμ για τα προγράμματα που έχουμε. Το συζήτησα χθε και με τον κύριο Σπίτλα, ε, όπως παραδείγματος χάρη ε, προφανώς συμβαίνει στο, στο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Οπότε είμαι υπέρ των καταποκοπήν ποσών και πρέπει να δείξουμε και εμπιστοσύνη στην υπευθυνότητα των κρατών μελών. γιατί χρηματο... συγχρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό ούτως ή άλλως αυτά τα ποσά. Η αλλω αυτα μου εμένα, η κύρια είναι, μέχρι στιγμής δεν το έχω εξετάσει λεπτομερώς, είναι πως λόγω της ε, παγκόσμιας αυτής όπως ξέρετε οικονομικής καταστροφής θα μπορούσαμε να καταθέσουμε μια τροπολογία για να έχουμε μια συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Το πρόβλημα μου είναι τώρα μην έχουμε δύο μέσα παράλληλα που θα λειτουργούν που θα πρέπει να ενισχύσουμε ταυτόχρονα. Να είμαστε πιο ακριβείς δηλαδή στους ορισμούς ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαν ευχαριστώ. Όπως σχεδόν πάντα σε αυτή τη ζωή με έπεισε η Καρνιγέννης, εγώ δεν θα υποβάλω τροπολογίες. Υπάρχει αρκετός έλεγχος και αυτό είναι σημαντικό, υπάρχει εγγύηση έλεγχου και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πράγματι είναι ουσιαστικό σε καιρό κρίσης ή εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν κάποια μέτρα κατάρτισης είναι ουσιαστικό σημείο και πράγματι παραμένει η ευθύνη στα κράτη-μέλη. Και κάτι άλλο που ανέφερε η κυρία Στάουνερ για τα, για τα Πράγματι μπορούν τα κράτη-μέλη να πούνε ναι εμείς καταπορεμάμε τη γραφειοκρατία και γίνεται αυτό με τα καταποκοπήν ποσά. Μπορούμε βεβαίως να καταργήσουμε τελείως τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινήσουμε από αυτό. Με έπεισαν οι δύο κυρίες. Ευχαριστώ. Δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, θα μιλήσω εγώ, να κάνω μια παρατήρηση. Ναι, κύριε Λέιντε, δεν σας είδα, συγγνώμη. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ε, μία σύντομη παρατήρηση είναι για να συμφωνήσω με τους ε, προαλήσαντες. Ε, κατά τύχη ε, έκα, συναντήθηκα με διάφορες ε, ενώσεις ε, στη Γαλλία που χρησιμοποιούν τα κονδύλια του ΕΚΤΕ για διάφορες δραστηριότητες. Τέλος πάντων. Ε, και συνάντησα διάφορες δυσκολίες. Ε, αλλά δυστυχώς σχετίζεται αυτό περισσότερο με την ε, διαχείριση των κονδυλίων σε γαλλικό επίπεδο και όχι σε ευρωπαϊκό. Πρώτον, καθυστερούν πάρα πολύ οι πληρωμές και οι σύνδεσμοι που δεν έχουν πολύ ρευστότητα σταματάνε τις δραστηριότητες τους όσο περιμένουν τα κονδύλια γιατί ζητάνε τις πληρωμές, αλλά το ίδιο και για τους εργαζόμενους, για τις ε, κοινωνικές εισφορές κτλ. Τη ζητάει βέβαια και η γαλλική κυβέρνηση, τέλος πάντων δεν έχουν λεφτά, οπότε σταματάνε ε, τις δραστηριότητες τους. Και άλλες πάλι ούτε καν το προσπαθούν, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαρτικά περίπλοκο το σύστημα και οι υπεύθυνοι δεν γνωρίζουν, δεν κατέχουν την κατάσταση και άρα τελικά παρετούνται. Ε, υπάρχει θέμα ταχύτητας, ε, καταβολής των πληρωμών και από, ε, σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και κατά τη γνώμη μου καλό θα ήταν να υπάρξει μια κατάρτιση και στους δημοσίους υπαλλήλους στα κράτη-μέλη και στα μέλη των ενώσεων, των συνδέσμων ε, για αυτή τη διαδικασία που είναι μεν εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά πραγματικά δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα πρακτικής εφαρμογής. Ωραία. Εγώ θέλω να υπερθεματίσω. Η αρμόδια αρχή στη Σουηδία, όπως είπε και ο κύριος Λέιντε και άλλοι, μα ενημερώνει ότι υπάρχουν πολλοί που παρετούνται, ε, πολλές ε, νόσεις που, σύνδεσμοι που θεωρούν ότι παρά είναι περίπλοκο το σύστημα. Εμείς ε, έχω, στη Σουηδία αναπτύχθηκε και δραστηριότητα παροχής συμβουλών, δηλαδή για να μαθαίνει κάποιος πόρους από το ΕΚΤ απευθύνεται σε συμβούλους για τον τρόπο για τις οδηγίες χρήσης, ας το πούμε Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποβάλει κανείς έτοιμα για κονδύλια. Ε, κονδύλια που όμως όλοι συμφωνούν επ' αυτού μπορούν, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οπότε ε, με τα νέα μέτρα θα μειωθεί η γραφειοκρατία και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούν οι εθνικές αρχές να βοηθήσουν στην πράξη της ενώσης ε, να χρησιμοποιούν, να υποβάλουν αιτήματα για κονδύλια. Δεν υπάρχει κανείς από την Επιτροπή, οπότε θα δώσω το λόγο λάθος έκανε ο Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή, λάθος μου τα είχαν πει, συγγνώμη, καλώς ορίσατε, σας δίνω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Λίγα πράγματα θα ήθελα να πω. Κατανοούμε τις ε, δυσκολίες ε, εφαρμογής όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και σε αυτή τη λογική κινούνται και οι τροποποιήσεις που προτείνουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι έτσι θα επιληθούν τα προβλήματα, ειδικά για τα μικρότερα έργα, τις μικρότερες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για τις οποίες θα υπάρξει σημαντική απλοποίηση. Θεωρώ ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης επειδή έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρά ποσά και άρα με πολύ μεγάλο αριθμό αποδείξεων και τιμολογίων. Κάτι που δημιουργεί δυσανάλογο γραφειοκρατικό άχθος σε σχέση με το ποσό των κονδυλίων. Ήδη από το πρώτο γύρο είχαμε την διάταξη που αφορούσε το άμεσο κόστος. Τώρα περνάμε και στα προκατακοπή ποσά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην κυρία Γέννης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για το ότι συμφωνούν μαζί μου και με την διαδικασία. Να αφαιρθώ με ευκαιρία την συζήτηση αυτή πως υπάρχουν κάποιες σκέψεις να έχουμε μια νέα αναπροσαρμογή ουσιαστική του περιεχομένου με ευκαιρία την κρίση και μιλάμε και για άλλα ταμεία. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό επόμενο βήμα και να ξαναδούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, επί της ουσίας στο ταμείο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να το ξαναδούμε. Όπως σας είπα αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ευχαριστώ για την συμφωνία σας.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 θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε το θέμα της ε, νωρίτερα. Κυρία Στάουνερ, έχετε εσείς επίσης κάτι για το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης μπορούμε να το δούμε σήμερα το πρωί. Συμφωνείτε? Ναι, πρέπει να ίσως να ενημερώσουμε τους σκιώδηγητές. Θα το δούμε. Και την ε, Κομισιόν. Ναι. Ίσως να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με το Ταμείο της ε, Παγκοσμιοποίησης, γιατί αυτό είναι ε, δική μας αρμοδιότητα. Ίσως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το απόγευμα. Ε, ίσως τώρα για την κυρία Μαδέρα να το δούμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη, πρώτη έκθεση της κυρίας Μαδέρα κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη, αρχές ενέργειες και μέσα. Γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ελευθεριών. Κυρία Μαντέρα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και σας ευχαριστώ για την προσπάθειά σας να κάνετε κάποιες χρήσιμες τροποποιήσεις στην ημερησιά διάταξη. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω τώρα τις δύο αυτές εκθέσεις γιατί αν τελειώσουμε γύρω θα μπορέσω να φύγω και για να συμμετέχω στην αποσχολή το του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Γάζα. Λοιπόν, η έκθεση για την κοινή πολιτική μετανάστευσης Έχουμε ήδη συζητήσει τη γνωμοδότηση Βεβαίως αυτή τη στιγμή βλέπουμε τη μετανάστευση στα πλαίσια της γενικής οικονομικής κρίσης. Αλλάζει λοιπόν η αντιμετώπιση μας και για τη μετανάστευση με βάση την υπάρχουσα οικονομική κρίση. Εγώ από την πλευρά μου Θεωρώ ότι μπόρεσα σε αυτή μου τη γνωμοδότηση να κρατήσω μία σαφή και συνεκτική γραμμή σε σχέση με παλαιότερες γνωμοδοτήσεις. Αναφέρω ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε δίκαιη και σωστή μεταχείριση όλων των μεταναστών. Γενικά μπορώ να συμφωνήσω με αρκετές τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι υπήρξαν προβλήματα στην Επιτροπή με το συγκεκριμένο σχέδιο γνωμοδότησης. Ορισμένες προτάσεις όμως θεωρώ ότι είναι υπερβολικά περιοριστικές περιορίζουν το εύρος των στόχων μας, εάν θέλετε. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι γενικά υπάρχει συνένεση επί της νομοδότησης. Θα ήθελα πάντως να λάβω μία-δύο διευκρινήσεις για κάποιες ε, τροπολογίες. Τροπολογία 20 της κυρίας Μωράν, για παράδειγμα. Όσον αφορά την ε, κατάρτιση και τις αρμοδιότητες ε, των τοπικών αρχών σε σχέση με την κατάρτιση δεν καταλαβαίνω αν το εννοεί ως παράδειγμα ή ως περιορισμό εδώ. Αν δείτε την τροπολογία θα μπορούσαμε να τη θεωρήσουμε ως περιοριστική για την αναζήτηση λύσεων που βασίζονται στον συντονισμό και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ε, παλαιότερες ε, αποφάσεις μας. Μήπως η κυρία Μωράν θα μπορούσε να μου διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί. Ευχαριστώ. Κυρία Ματέιρα, η κυρία Μωράν δυστυχώς απουσιάζει. Μπορούν όμως οι υπόλοιποι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο. Ζητάει κάποιος το λόγο. Η Επιτροπή. Όχι. Κυρία Παναγιωτοπούλου. Ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την κυρία Μαδέρα για την ε, ευαισθησία της ε, στο θέμα που φαίνεται μέσα από το κείμενο που έχει δώσει. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα με την κυρία Μωράν θα πρέπει να λυθεί με την ίδια, ίσως να πρόκειται και για δυσκολία της μετάφρασης. Θα ήθελα όμως να παρατηρήσω ότι πολλές τροπολογίες κυρίας Μαδέρα στέκονται στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ε, επίπεδο. Μια μικρή παρατήρηση ότι είναι κάπως ε, διάσπαρτες και ε, πολύ τονισμένες οι τροπολογίες που αφορούν την εκπαίδευση και την πολιτιστική διάσταση του προβλήματος. Κατά τα άλλα νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μαζί καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πανακιατοπούλου. Κάποιος άλλος θέλει να σχολιάσει. Όχι. Κυρία Ματέιρα, θέλετε να συνοψίσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ αγαπητοί συνάδελφοι θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές συμφωνούμε Δεν ξέρω αν το θέμα που ανέφερα με την κυρία Μωράν είναι θέμα μετάφρασης, αλλά ακόμη και αν όχι σίγουρα νομίζω ότι συμφωνούμε επί της πρότασης και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία πρόταση για την πολιτική μετανάστευση που θα σέβεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του θέματος αυτό. Στις 2 Μαρτίου θα έχουμε την ψηφοφορία επί του θέματος. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση της κυρίας Παναγιωτοπούλου που αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι ε, τροπολογίες, 52 ε, τροπολογίες υποβλήθηκαν στην έκθεση για την οποία έχουμε ξανασυζητήσει. Το κύριο θέμα της... Το δεν θα ε, μιλήσω για την ίδια την πρόταση γιατί έχουμε ξανασυζητήσει. Θα μιλήσω ειδικά για τις τροπολογίες. Η τροπολογία 9 ε, που απορρίπτει την πρόταση ε, την αφήνω στην κρίση των συναδέλφων. Νομίζω ότι αφού διαπιστώθηκαν δυσκολίες στην εφαρμογή ε, αυτό είναι ε, νομίζω από όλους αποδεκτό και φαίνεται και από την ε, έκθεση της Επιτροπής. Μπορεί η έκθεση της Επιτροπής να μην μας αφήνει να δούμε πολλά πράγματα, ίσως από έλλειψη αποστολή στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι μια έκθεση που μας ικανοποιεί όμως το ότι ε, δεν είναι τέλεια στην εφαρμογή της η οδηγία του 2002 είναι από όλους αποδεκτό. Αν λοιπόν απορρίψουμε την πρόταση της ε, Επιτροπής ε, είναι σαν να κλείνουμε το διάλογο. Γι' αυτό και η τροπολογία 9 που απορρίπτει την πρόταση δεν νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση για να βελτιώσουμε την πρόταση και όχι να την απορρίψουμε. Ε, η άλλη τροπολογία για την ένταξη των αυτοαπασχολουμένων είναι η βασική, ε, μια, ένας από τους βασικούς άξονες ε, της συζήτησης. νομίζω ότι και εκεί υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις και χρειάζεται πραγματικά διάλογος σε βάθος και όχι ε, ανάταση κάποιας κομματικής ε, σημαίας υποστηριζόμενης από ε, συμφέροντα ομάδων. Να συζητήσουμε στο βάθος τι είναι ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας αληθινός αυτοαπασχολούμενος και τι είναι ένας ε, κατά τον τύπο από απασχολούμενος και να βρούμε τρόπους να εξαιρέσουμε αυτούς που είναι κατά τον τύπο αυτοαπασχολούμενοι αλλά να μην θίξουμε αυτούς που είναι... Ε, τώρα νομίζω ότι δεν πρέπει να συνεχίσω. Τι να κάνω. Ε, ε, να μην Εδώ γίνεται συζήτηση ή δεν γίνεται κυρία Πρόεδρε. Μπορείτε να με πληροφορήσετε. Uh, ναι, με συγχωρείτε για τα σημερινά πράγματα. Είναι κάπως ε, μπερδεμένα τα πράγματα. Με συγχωρείτε για την κατάσταση σήμερα το πρωί. Στίβεν Χιούζ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων έχει θεμελιώδη σημασία. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν τελείωσα. ε, ε, μετέβωσε κουτάκι. Okay, excuse me. Go on then. Με συγχωρείτε, συνεχίστε τότε. Some, sorry, it was some confusing. Με συγχωρείτε, ήταν λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Okay. Τα ακουστικά με το yeah. να I, I speak, yes. Ναι, επικράτησε μία μικρή σύγχυση γιατί συζητούσαμε τα, τα των εγγύων ε, γυναικών. Ε. Εντάξει, υπήρξε τώρα μία μικρή σύγχυση, κάποιοι συναδελφοί παραπονιούνται, λένε πως ε, θέλουν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να έρθει οπωσδήποτε αυτό το θέμα το απόγευμα. Οπότε μπορούμε, πρέπει ίσως να ξαναλλάξουμε την ενημερίσια διάταξη. Πάντα είναι προβληματικό αυτό και, δύσκολο. Γιατί κάποιοι περίμεναν ε, να, έρθει αργότερα αυτό το θέμα και ενδιαφέρονταν. Ε, με συγχωρείτε κύριε Παναγιωτοπούλου, έχετε τον λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, με το να μην φοράτε τα ακουστικά σας, δεν παρακολουθείτε τη συζήτηση. Εγώ δεν είχα τελειώσει την ε, ε, ε, συζήτηση των τροπολογιών και δώσατε το λόγο στον κύριο Χιούτς ενώ εγώ δεν είχα τελειώσει τη συζήτηση. Έλεγα λοιπόν ότι η τροπολογία 12 με την ένταξη των αυταπασχολούμενων θέλει περισσότερη συζήτηση γιατί νομίζω ότι κανένας δεν είναι κατά της δημιουργίας ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υγιών επιχειρήσεων που βοηθούν τον ε, υγιή ανταγωνισμό αντίθετα όλοι θέλουμε να πατάξουμε φαινόμενα νόθευσης του ανταγωνισμού από ψεύτικους ε, αυτοαπασχολούμενους. είναι λοιπόν προς το συμφέρον των εργαζομένων να συνεχίσουμε να συζητούμε και να βρούμε ένα τρόπο ε, που θα αποκλείει τους ε, ε, απασχολούμενους και θα βοηθάει τους εργαζόμενους να έχουν τα δικαιώματά τους. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ στην εξαίρεση κάθε συζήτησης που αφορά το χρόνο και τις συνθήκες οδήγησης οι οποίες καλύπτονται από τον κανονισμό ε, τον ε, ενεργεία, τον ενισχύει ε, κανονισμό. Απορώ γιατί υπάρχουν τροπολογίες που φέρνουν τον παλιό κανονισμό μέσα στην πρόταση. Απορώ γιατί υπάρχουν τροπολογίες που φέρνουν την παλιά οδηγία του 1993 μέσα στην πρόταση. Θα ήθελα εξηγήσει επ' αυτού. και πιστεύω ότι η διαγραφή της ε, δυνατότητας ε, των κρατών μελών να προειδοποιούν τους οδηγούς για τις κακές συνθήκες θα μπορούσε να βελτιωθεί και να αποτελέσει ε, όχι μια συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων αλλά μια, ένα κάλεσμα προς τα κράτη-μέλη μιλώ ας πούμε για την τροπολογία 14 πως θα μπορούσε να βελτιωθεί ένα κάλεσμα προς τα κράτη-μέλη αυτά κατά τις δικές τους συνήθειες και ε, με αποτελεσματικό τρόπο να συμπεριλάβουν ή να μην συμπεριλάβουν κατηγορίες που θεωρούν κρίσιμες ε, πιθανότατα και την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων. Ε, και από αυτού θα ήθελα την μαρτυρία του κυρίου Χιούτς αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου η χώρα του συμπεριλαμβάνει τους αυτοαπασχολούμενους ε, ε, στην νομοθεσία ε, άλλες χώρες όμως έχουν δυσκολία να το πράξουν. επειδή είναι λοιπόν πολλές οι παραδόσεις στα 27 κράτη μέλη θα πρέπει να έχουμε ελαστικότητα και να κάνουμε μια οδηγία που θα μπορούν να την εφαρμόσουν όλοι και που δεν θα κρύβονται πίσω από αυτήν για να νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Ε, είμαι πρόθυμη λοιπόν να συζητήσουμε, άλλωστε έχουμε και το απόγευμα μία συνάντηση, ε, να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ε, ένα αποτέλεσμα θετικό για τους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους αφορά η οδηγία και πιστεύω ότι τους εργαζόμενους μόνο μπορούν να ελέγξουν οι ελεγκτές της εφαρμογής αυτής της οδηγίας όποιοι και να είναι από κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ κυρία Παναγιωτοπούλου. Στίβεν Χιούς και μετά Λέιντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Εγώ πρώτο είδα αυτή την έκθεση το, το, 2001-2002 όταν αποφασίσαμε να επεκτείνουμε τις οδικές μεταφορές στις οδικές μεταφορές το ζήτημα του χρόνου εργασίας και το σκεφτήκαμε σοβαρά το θέμα των αυτοαπασχολουμένων και την εξαιρεσή τους. Δεν είναι πολιτικό το ζήτημα, είναι πολύ ουσιαστικό. Τότε η Κομισιόν ήταν σαφής πως ε, έπρεπε να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Γι' αυτό χρησιμοποιούσαμε και μία ε, νομική βάση και ασφάλειας και υγιεινή συνεργασία και επιχειρησιακής ασφάλειας. Δεν ξέρω εάν ε, μελέτησε κανείς τη μελέτη που η Κομισιόν θα έπρεπε να είχε υποβάλει δύο χρόνια πριν για την συμπερίληψη ή όχι των αυτοαπασχολούμενων. Εν πάση περιπτώσει Πέρσι τον, τον Μάιο βγήκε η έκθεση αντί για πριν από δύο χρόνια. Εάν τη διαβάσετε θα δείτε πως υπάρχουν παντού σοβαρά επιχειρήματα για την συμπερίληψη των αυτοαπασχολημένων και ένα-δύο επιχειρήματα για την εξαίρεσή τους. Να σας αναφέρω μόνο ένα μικρό τμήμα της μελέτης. Λέει στην αρχική της ε, πρόταση και κατά διάρκεια της συζήτησης η Κομισιόν πρότεινε τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολημένων για πολλούς λόγους. Πρώτον, για να είμαστε συνεπείς με την σχετική οδηγία που δεν κάνει διάκριση μεταξύ των οδηγών. Δεύτερον, για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός ενός πολύ ανταγωνιστικού κλάδου με το να ορίζονται μετά όλοι οι οδηγοί ως αυτοαπασχολούμενοι. Τρίτον, για να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός που μόλις ανέφερε η συγκήτρια άλλωστε. Και Τέταρτον, για να υπάρχει οδική ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά, παρά μόνο η στάση της Κομισιόν. Και δεν βασίζεται στα στοιχεία, γιατί αν διαβάσετε τη μελέτη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Κουρασμένος αυτοαπασχολούμενος είναι επικίνδυνος ε, και για τον εαυτό του και για τους ε, υπόλοιπους. Δεν θα πρέπει να να αναρωτιόμαστε όταν βλέπουμε μια ανταλίκα απέναντί μας στο δρόμο εάν αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοαπασχολούμενος και δεν έχει κοιμηθεί και οδηγά 72 ώρες ή αν έχει ξεκουραστεί κανονικά. Γιατί πραγματικά εδώ πέρα ο καμισμός αυτός όπως προτείνεται θα επιτρέψει το να οδηγάνε οι αυτοαπασχολούμενοι 87 ώρες τη βδομάδα. Το αποτέλεσμα λοιπόν των δικών μου τροπολογιών είναι να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και ζητώ από την Επιτροπή να το υποστηρίξει. Διαβάστε σας παρακαλώ τη μελέτη. Το έγγραφο είναι COM 2007-266. Σας παρακαλώ διαβάστε τη μελέτη και ελάτε μετά να μου πείτε πώς πρέπει να εξαιρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Νομίζω είπε επίσης η γήτρια πως πρέπει να βρούμε έναν ορισμό για τους όντως αυτοαπασχολούμενους και τους ψεύδο αυτοαπασχολούμενους. Κοιτάξτε, ο ορισμός αυτός μας απασχόλησε πολύ το 2007. Είδαμε τους υπάρχοντες κανόνες στα κράτη-μέλη, το πώς ορίζουν τον αυτοαπασχολούμενο κτλ. Είναι πολύ σοβαρά κριτήρια που αν εφαρμοστούν σωστά θα βρουν πράγματι τους όντως αυτοαπασχολούμενους και αυτούς που στην πραγματικότητα από έναν εργοδότη εξαρτώνται. Νομίζω το έχουμε δει λοιπόν αυτό και στην αρχική οδηγία είδαμε το ζήτημα των διοικητικών ε, εργασιών για τους αυτοαπασχολούμενους ε, το... ξεκαθαρίσαν που δεν συμπεριλαμβάνεται αυτό ε, στον χρόνο εργασίας των οδηγών γιατί προφανώς δεν μπορεί να το επιτηρήσει κανείς οπότε αυτό υπάρχει ήδη στην αρχική οδηγία οπότε έχει σχεδιαστεί ήδη η οδηγία για να συμπεριληφθούν εύκολα οι αυτοαποσχολούμενοι. Πρέπει νομίζω να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν γιατί δεν είναι ειλικρινής με το Κοινοβούλιο εδώ πέρα. Έχουν, έχει μετατοπιστεί η θέση τους και δεν δικαιολογείται αυτό από τίποτα από αυτά τα οποία διάβασα. Είναι νομίζω κάτι το οποίο Φθέτει, ένα την καλή συνεργασία μας με την Κομισιόν στη διαδικασία της ε, συνδιαλλαγής και είναι επέσχυντο. Αλλιώς, ειλικρινά, δεν τους χρειαζόμαστε στη συνδιαλλαγή. Καλύτερα να μιλάμε απευθείας με το Συμβούλιο. Και ελπίζω να το μεταφέρουν αυτό το μήνυμα. Η θέση μου τώρα είναι σαφής. Να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν, να κάνουν μια σωστή μελέτη και να φέρουν μια πρόταση να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι. Εάν όχι, να υποστηρίξουμε τις δικές μου τροπολογίε που έχουν το ίδιο αποτέλεσμα την συμπεριλήψη των αυτοαπασχολούμενων. Ευχαριστώ Καϊντέ και, Κρέιντερ και Κρέμερ μετά έχουμε στον κατάλογο. Λοιπόν, η πρόθεση η δική μου ήταν το θέμα της κυρίας Μαντέιρα να πάει την απογευματινή συνεδρίαση αλλά άλλοι συνάδελφοι παραπονέθηκαν λέγοντας πως περίμεναν να συζητηθεί αυτό το πράγμα το απόγευμα και θα ερχόταν το απόγευμα αυτοί να το συζητήσουν και πάντα υπάρχουν τέτοια προβλήματα όταν αλλάζει η μερίσια διάταξη οπότε δεν θα αλλάξει το ε, σημείο σας αυτό θα συζητηθεί το απόγευμα όπως είχε προγραμματιστεί υπήρχαν ε, Κάποιοι λόγοι δεν ψήφισαν την έκθεση Μπραγκέτο, είχαμε λίγο χρόνο παραπάνω. Λυπάμαι, κανονικά δεν θα ήθελα να αλλάξω την μερίσια διάταξη, αλλά τέλος πάντων ε, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Η κυρία Μαντέιρα Πρόεδρε, όπως σας είπα, Λυπάμαι ε, που δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μου, τα αιτήματα που έκανα την περασμένη εβδομάδα και τώρα ανακύπτουν εκ νέου για την τροποποίηση δηλαδή, της ημερήσιας διάταξης. Από όσο ξέρω, όταν υπάρχει, ε, όταν έγινε το αίτημα δεν αναφέρθηκε ότι υπάρχει κάποιο κόλλημα. Τέλο πάντων, δημιουργείται προηγούμενο τώρα και λυπάμαι. Λυπάμαι ε, που ε, έχει γίνει λίγο τσίρκο εδώ. Δηλαδή, εντάξει, ε, υπάρχουν οι επισκέπτες, τους σέβομαι, αλλά έχουμε και μία ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, για να προβάλλουμε επικοινωνιακά την εικόνα μας, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Λυπάμαι. will not floor. Uh, fru Κυρία Μαντέιρα, την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει ότι θα το μεταφέρουμε την Τρίτη και εγώ το αρνήθηκα ως Πρόεδρος για τον απλό λόγο ότι εχθές ε, είχαμε γεμάτη μέση διάταξη με γνωμοδοτήσεις που θα ψηφίζαμε σήμερα και ε, στις 6 έπρεπε να τα πούμε στους συντονιστές για την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Ήταν εντελώς διαφορετικά το θέμα και γι' αυτό το αρνήθηκα και εμένω στη θέση μου. Ήταν αδύνατον εχθές. Τώρα τι γίνεται σήμερα. Επειδή ε, υπήρχαν ε, οι ψηφοφορίες, σκέφτηκα να το αναβάλουμε το απόγευμα, αλλά αυτό είναι ξεχωριστό θέμα. Και δεν είχα πρόβλημα γιατί υπήρχε περιθώριο. Ε, και ε, είπαν τα μέλη της Επιτροπής ότι ήθελαν να παραστούν στη συζήτηση εφόσον έχει προβλεφθεί για το απόγευμα και γι' αυτό έκρινα έτσι, αλλά είναι δύο διακριτά ζητήματα. Ένα ήταν ότι θα πήγαινε την Τρίτη το θέμα, αλλά αυτό ήταν αδύνατον δεδομένης ημερησίας διάταξης. Τέλος πάντων θα το συζητήσουμε το απόγευμα. Θα ακολουθήσουμε την αρχική ημερήσια διάταξη. Λυπάμαι. Ε, αναγκάστηκα να λάβω αυτή την απόφαση. Σας ενημερώνω ότι θα ακολουθήσουμε λοιπόν την ε, ημερήσια διάταξη όπως ακριβώς την είχαμε σχεδιάσει. Ο κύριος Λέιντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Επειδή τελικά θα χάσουμε το χρόνο που κερδίσαμε από την μη ψήφιση της έκθεσης Πραγκέτ, θα ήθελα να επανέλθω στη συζήτηση της έκθεσης και να πω κάποια πράγματα πολύ σύντομα. Καταρχάς, το πιο σημαντικό θέμα για εμάς είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και όσων κυκλοφορούν στους δρόμους. Είναι δύο πολύ βασικά θέματα. Δεν θέλω να αλλάξει το νομικό καθεστώς των οδηγών φορτηγών. Είτε είναι μισθωτοί είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, τα προβλήματα ασφάλειας έχουν την ίδια φύση. Και οι κίνδυνοι που υπάρχουν αν δουλεύουν υπερβολικά αν κυκλοφορούν ε, πολλές ώρες τη νύχτα κτλ. παραμένουν τα ίδια. Η Κομισιόν δεν ξέρω αν ακάλυψε λόγους ε, για να αλλάξει το καθεστώς, αλλά αν υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος θα πρέπει να μας το πει. Βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι πραγματικά αυτοαποσχολούμενοι. Νομίζω ότι αυτή η απλούστευση δεν είναι κατανοητή. Επίσης, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των αυτοαποσχολούμενων εργαζόμενων και των μετακινούμενων εργαζόμενων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι αυτό αυτοαπασχολούμενος, αλλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για μετακινούμενο εργαζόμενο. Γιατί στη Γαλλία τουλάχιστον μετακινούμενος είναι κάποιος ο οποίος μετακινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Ναι, όλοι οι οδηγοί μετακινούνται κατά αυτή την έννοια. Εγώ θεωρώ ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Και αν διαφωνεί η Κομισιόν πρέπει να μας εξηγήσει ακριβώς γιατί τώρα αποφάσισε να τους εξαιρέσει. Θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στην Κομισιόν. Η κυρία Μαντέιρα παρακαλώ. Διαδικαστικό. Ε, συγγνώμη, ε, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Μετά τις ε, διευκρινήσεις που μου δώσατε και τρέφω σεβασμό για σας, απλά θέλω να τονίσω ότι σε επόμενες συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η μερίσια διάταξη, δηλαδή ποτέ δεν θα πρέπει να τροποποιείται τη μερίσια διάταξη, ακόμη και ένα μέλος της Επιτροπής να αντιτάσσεται, όχι μια πολιτική ομάδα, ακόμη και ένα μέλος της Επιτροπής. Ε, να αντιτάσσεται. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Ε, και τώρα σε αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει στην Επιτροπή μας θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ποια είναι η μυρίσια διάδεξη από το 24 ως το 31. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι όπως είναι στους φακέλους μας. Απλά τώρα για να το διευκρινίσετε και αυτό γιατί μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω τι αποφασίσατε. Vi lag. Ναι, ναι, θα ακολουθήσουμε αυτή την μέση διάταξη που έχετε. Θα συνεχίσουμε με την κοινή συζήτηση για τις νομοδοτήσεις ε, της κυρίας Λάμπερτ και του κυρίου Κρέμερς ε, και μετά θα ακολουθήσουμε την ημερήσια διάταξη όπως ήταν ε, για το απόγευμα, τη δική σας έκθεση, τη μελέτη, την έκθεση της κυρίας Τάουνερ και τα λοιπά. Ο κύριος Κρέμερς και η κυρία Φικυρίδα ακολουθούν. Ε, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορεί να είμαι πολύ σύντομος γιατί επί της αρχής ε, μπορώ να συμφωνήσω με τον ε, Steve Hughes. Πρέπει όμως να αναφέρω κάτι εδώ γιατί δεν φαίνεται τόσο η διαφορά μεταξύ αυτοαπασχολούμενου και ψευδοαπασχολούμενου. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη μελέτη που είχε γίνει από το καθηγητή Μπορούντι και που αφορούσε τις ανάγκες τις νομικές τότε είχε αναφερθεί ότι πρέπει να υπάρξει ένα σαφής ορισμός του τι εννοούμε με τον όρο αυτοαπασχολούμενος προκειμένου να μην γίνεται κατάχρηση του όρου. Εγώ θα συμφωνούσα με μία τέτοια ξεχωριστή νομοθεσία αλλά δεν θεωρώ ότι εντάσσεται σε αυτό το φάκελο αυτό το θέμα δεν μπορεί να επιληφθεί σε ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να είναι μια ξεχωριστή ατζέντα. Ευχαριστούμε η κυρία Φιγκυρέντο και η κυρία Φανλάνγκεν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε αυτή τη συζήτηση πριν από λίγα χρόνια στην Επιτροπή και νομίζω ότι ε, καρκινοβατούμε και επαναρχόμαστε σε αυτό που είχαμε αποφασίσει. Είχαμε πει ότι θα συμπεριλαμβάναμε τους ανεξάρτητους επαγγελματίες. Μα, ε, το είχαμε συζητήσει επί μακρόν το θέμα. Και είχαμε πει ότι ε, έπρεπε να συμπεριληφθούν στην οδηγία οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Η Επιτροπή και άλλοι είπαν ότι άμα είναι να γίνει έτσι χρειάζεται μεταβατική περίοδος και άρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό. Και σήμερα δηλαδή πανερχόμαστε, ανακαλούμε αυτό που αποφασίσαμε ή θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση σαν να μην είχε γίνει. Συγγνώμη, δεν είναι σωστό αυτό ούτε καν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω, εντάξει, μάλλον δεν είναι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι ορθή αυτή η πρόταση λοιπόν που μας κάνει η Επιτροπή και γι' αυτό προτείνουμε να αντιταχθούμε σε αυτή την πρόταση υπαναχώρησης ανάκλησης ε, του, της απόφασης του Κοινοβουλίου. Για τότε το Κοινοβούλιο, σας λέω, είχε δεχτεί ε, την πρόταση της Επιτροπής για να ρυθμιστεί ε, αυτό το ζήτημα και τώρα τι, ε, τα αμφισβητούμε όλα και ανακαλούμε την απόφασή μας, δεν καταλαβαίνω, δεν, μπορούμε, δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις μας. Ξαναλέω, το είχαμε συζητήσει το θέμα, το είχαμε εγκρίνει, είχαμε αφασίσει τότε για αυτό το θέμα. Πρέπει να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να λήξει αυτή η κατάσταση των ψεύδο αυτοαπασχολούμενων για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί πρόκειται για τα δικαιώματα όλων των απλών ανθρώπων που ε, κυκλοφορούν δεν υπάρχουν, υπάρχει ασφάλεια, χρόνος, κατοχυρωμένος χρόνος ανάπαυσης λοιπά. Μα άμα συμβαίνει αυτό, όλοι οι απλοί άνθρωποι θα υποφέρουν, θα πληγούν από αυτό. Λυπάμαι που μας προτείνει κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Φανλάνκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ότι είναι παράλογο να κάνουμε διάκριση μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων όταν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η οδική ασφάλεια και η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων. Βεβαίως θέλουμε να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός, γι' αυτό όμως πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλους. Φαίνεται ότι έχει χάσει η συγγήτρια την έκθεση του Οκτωβρίου, όπου με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε στην Ολομέλεια ότι θέλουμε να συμπεριληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην οδηγία. Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια στάση παντού και εδώ. Και μία ερώτηση προς τον κύριο Χιούς. Ναι, μεν ε, οι περισσότεροι μας συμφωνούμε, αλλά πρέπει να πείσουμε και τους συγητές. Οπότε, ως μέλος ε, του Κοινοβουλίου Αναρωτιέμαι, είναι καλύτερα να απορρίψουμε την πρόταση ή να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν, συμπεριλαμβάνοντας τους αυτοαπασχολούμενους, έτσι ώστε να καταφέρουμε πράγματι αυτό που επιθυμούμε. Μήπως μπορείς να μου απαντήσεις, ε, Στίβεν, ε, ποια θα είναι η στρατηγική σου ή μάλλον ποια είναι η στρατηγική σου όταν προτείνεις την απόρριψη. Ευχαριστώ. Eh, ε, τώρα κάνετε ερωτήσει σε κάποιον που δεν είναι εισηγητή, οπότε δεν μπορεί να βρείτε έναν τρόπο να το ρυθμίσετε για να συνεχίσουμε εμεί τη, συζή... τη, συζήτηση. Συγγνώμη, η κυρία Τομασεύσκα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για εμένα το θέμα του θέμη του ανταγωνισμού είναι μικρή σημασία σε σχέση με το σημαντικότατο θέμα της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζουμε ότι ατυχήματα στο δρόμο συμβαίνουν συνεχώς είτε κάποιος είναι οδηγός είτε όχι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος είτε όχι. Το ζητούμενο εδώ είναι να μπορούν οι οδηγοί να ανταποκρίνονται άμεσα στην οποιαδήποτε μεταβολή, στο οτιδήποτε τυχαίο συμβεί κάποια στιγμή στο δρόμο. Ίσως θα έπρεπε να προτιμήσουμε τη λύση της κυρίας Βαν Λάνκερ ή να συμπεριλάβουμε κάποιες διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι εργαζόμενοι του τομέα, είτε είναι μισθωτοί είτε όχι, θα πρέπει να οργανώνουν το χρόνο εργασίας τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελοχιστοποιούνται τα οδικά ατυχήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει άλλο στον κατάλογο μιλητών. Θέλω να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε πάρα πολλές ε, διαφορετικές απόψεις. Σας ακούσουμε τώρα τον κύριο Σμίτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ ξανά στο βασικό ζήτημα, τι θα γίνει δηλαδή με τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. Και ποιους λόγους έχει η Κομισιόν για να προτείνει την εξαίρεσή τους. Θα ήθελα να αναφέρω τρεις λόγους να έχετε υπόψη σας. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση πριν από 11 χρόνια ήταν θεμελιωδώς διαφορετική από τη σημερινή όσον αφορά τους χρόνους οδήγησης και ξεκούρασης από το 2007. Έχουμε αυστηρές διατάξεις που ελέγχονται κιόλας για τον χρόνο οδήγησης και αφορούν όλους τους οδηγούς ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης και κατά μέσο όρο ένας οδηγός δεν μπορεί να οδηγά τη βδομάδα πάνω από 45 ώρες. Κάθε οδηγός. Πριν από 11 χρόνια δυστυχώς η κατάσταση ήταν τόσο διαφορετική που μπορούσε να οδηγεί κάποιος 80 ώρες τη βδομάδα που βεβαίως είναι μια τελείως απαράδεκτη κατάσταση για την οδική ασφάλεια. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ πως ε, το μεγαλύτερο κομμάτι της απασχόλησης και των υπαλλήλων και των αυτοαπασχολουμένων είναι η οδήγηση. Και αυτό το έχουμε ρυθμίσει πάρα πολύ καλά πλέον μέσω, τα του, το, μέσω των του χρόνου οδήγησης και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε εδώ πέρα μέσω του χρόνου εργασίας. Επίσης, το να επεκτείνουμε κάτι για τον χρόνο εργασίας στους ε, αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή κατ' ουσίαν στους επιχειρηματίες, είναι πρωτοφανές. Πουθενά δεν ισχύει αυτό. Πράγματι και οι αυτοαπασχολούμενοι κατά κανόνα έχουν την τάση να εργάζονται μέρος του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε αυτή την επιχειρηματική ελευθερία να την περιορίσει. Και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα είναι βεβαίω το ζήτημα της εφαρμογής. Κατά τη διάρκεια των μελετών μας εξετάσαμε εις βάθος αυτό το ζήτημα και φαίνεται αυτό και στην έκθεση του 2007 της Κομισιόν. Η εφαρμογή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα ήδη της υπάρξης οδηγίας. Φανταστείτε να επεκταθεί και στους αυτοαπασχολούμενους. Δεν θα εφαρμόζεται στην πράξη. Εκτός εάν γυρίσουμε στις ε, αρχές του Όργουελ και βάλουμε ένα μεγάλο αδερφό και καταγράφει κάθε κίνηση του καθενός διάφανα έτσι να τα βλέπουν όλα οι αρχές. Αυτοί λοιπόν οι τρεις λόγοι θεωρώ πως συνηγορούν στο να μην επεκτείνουμε εδώ πέρα την αρχή αυτή και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί μέχρι κεραίαση υπάρχουσα νομοθεσία, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει. Οπότε, στηρίζουμε πλήρως ε, την ε, εισηγήτρια όλες οι αλλαγές που υπάρχουν και έχουν στόχο να βελτιώσουν τον έλεγχο είναι πολύ σωστές. Στόχος πρέπει να είναι επίσης οι παραβιάσεις οδηγίας να έχουν επαρκείς κυρώσεις, αλλά είμαστε ρητός κατά της επέκτασης τώρα αυτής της οδηγίας τους αυτοαπασχολούμενους. Και να δημιουργήσουμε δηλαδή έτσι ένα κείμενο το οποίο δεν θα έχει αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Τέλος, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας που συνεχώς αναφέρεται και είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα για την Κομισιόν. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε εις βάρος της οδικής ασφάλειας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Όπως σας είπα, οι χρόνοι οδήγησης και ξεκούρασης έχουν ξεκαθαρίσει ήδη από το 2007. Σε αυτό προστίθεται πως οπωσδήποτε η κούραση είναι σημαντικός παράγοντας για τα ατυχήματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού προέρχεται η κούραση δεν είναι οπωσδήποτε το, από το ότι εργάζονται οι ε, επιχειρηματίες, είναι θέμα ποιότητας του ύπνου, της ποσότητας του ύπνου και του στρες και του βιολογικού ε, ρολογιού. Και εκεί πέρα έχουμε ε, οπωσδήποτε περισσότερες προβλήματα με τους υπαλλήλους εταιριών που ε, ε, αντιμετωπίζουν νομερή πίεση από τις εταιρείε τους αλλά οι αυτοαπασχολούμενοι τουλάχιστον δεν θεωρώ πως ε, τους αγγίζει ιδιαίτερο αυτό το πρόβλημα οπότε σας παρακαλώ να δείτε με αυτό το μάτι την πρόταση της Κομισιόν όπως προτείνει και η συγκεκριμένη Ευχαριστώ. Ο Στίβεν Κιούς έχει ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό. Κατόπιν μπορούμε να περάσουμε στο θέμα της κυρίας Αν Φανλάνκεν. Για να απαντήσει ίσως την κυρία Αν Φανλάνκεν και μετά ακούσουμε την εισηγήτρια. Κύριε Στίβεν Χιούς, διαδικαστικό απλά ενημερωτικό προς την Επιτροπή. Λέει η Επιτροπή ότι αν το παρατείνουμε αυτού του αυτοαπασχολούμενου, ε, θα παραβιάσουμε την ε, παράδοση. Για πρώτη φορά δεν αληθεύει αυτό. Ας δει τη σχετική οδηγία για ε, την κινητικότητα των εργαζομένων θα δει ότι υπάρχει προηγούμενο και ούτως ή άλλως έχουμε και το ΔΕΚ. Μετά το, την έγκριση το 2002 η Φινλανδία και η Ισπανία, δεν κάνω λάθος, παρέμβησαν το θέμα ενώπιον του δικαστηρίου για το θέμα των αυτοαπασχολουμένων και απερίφθη το αίτημά τους από το ΔΕΚ. Είναι ψευδό το επιχείρημα, μην το επικαλείστε ε, και να είστε ειλικρινείς ενώπιον της Επιτροπής μας. Ε, και ακριβώς επειδή δεν είναι ειλικρινή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το απορρίψουμε και να τους παραπέμψουμε σε αυτά που είχαν αποφασιστεί το 2001 και 2002. Αν δεν ε, αυτό στην Ολομέλη είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποβάλουμε τις τροπολογίες και να τροποποιηθεί αναλόγως το κείμενο. Ευχαριστώ. Η, θα ακούσουμε την εισηγήτρια. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Η κυρία Παναγιωτοπούλου θα συνοψίσει τη συζήτηση. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι η συζήτηση δεν είχε ποιότητα. Ήταν σαν να πεζόταν δύο θεατρικά έργα το έργο της κυρίας ε, Μαντέιρα και ο χρόνος εργασίας των οδηγών και βλέπαμε μία πράξη του έργου της κυρίας Μαντέιρα και μία πράξη του έργου των οδηγών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση είχε ποιότητα. Ύστερα ε, να αρθούμε στην ουσία ξεκαθαρίστηκε το θέμα ότι δεν αφορά την οδήγηση, δεν αφορά ε, καθόλου την κούραση που προέρχεται από την οδήγηση η οποία ρυθμίζεται από τον κανονισμό. Άρα δεν πρέπει να βάζουμε μέσα ούτε το θέμα της αμοιβή που ε, δεν το αφορά η ε, πρόταση αυτή ούτε το θέμα της οδήγησης. Ε, κάθε φορά λοιπόν που στοχεύουμε στο συνέστημα προκαλώντας τον τρόμο και τον ίκτο για τους πεζούς από τον κίνδυνο των οδηγών που είναι κουρασμένοι κάνουμε λάθος. εδώ πρόκειται για μια οδηγία που έχει άλλο στόχο. νομίζω ότι ο κύριος είχε απόλυτο δίκιο να λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της κούρασης των οποιονδήποτε οδηγών ξεχωριστά ε, ε, όπως έχουμε τα αλκοτέστ για τους ε, οδηγούς που έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διασκεδάζουν αλλά οφείλουν να μην είναι μεθυσμένοι έτσι πρέπει να έχουμε κάποιο τρόπο να βρούμε και την κούραση και νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιοι τρόποι να μετρηθεί η κούραση του οποιοδήποτε οποιοδήποτε οδηγού όχι όμως του επιχειρηματία μόνο ε, και του εργαζόμενου μόνο. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να νοθεύσουμε την έννοια του εργαζόμενου και την έννοια του επιχειρηματία. εδώ έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις και βέβαια θέλουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. απ' την άλλη πάλι δεν θέλουμε να μπλέξουμε μέσα την έννοια του επιχειρηματία ως προς την ε, ε, αυτονομία του ως επιχειρηματία. Νομίζω ότι όλοι μας είμαστε υπέρ του να υπάρχουν υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν λοιπόν δεν αφήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις χωρίς εμπόδια ε, ως προς ε, την διάθεση του χρόνου τους, άλλο η κούραση. Η διάθεση του χρόνου όμως δεν μπορεί να οριστεί από μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν, είμαστε, ε, ε, δεν έχουμε δικαίωμα να επέμβουμε στην ιδιωτική ζωή ενός επιχειρηματία. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη να ελέγξουμε το χρόνο εργασίας ενός εργαζόμενου. Έχουμε ευθύνη ο εργαζόμενος να μην ε, ε, ε, του γίνεται κατάχρηση. Νομίζω ότι μπορούμε να προτείνουμε κάποιους άλλους τρόπους να ελέγξουμε την κούραση του οποιοδήποτε οδηγού είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι εργαζόμενος ε, θα ήθελα όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι δυνατόν να δευτερολογήσει για να μας μιλήσει για τη δικαστική απόφαση την οποία αναφέρει ο κύριος Χιούς και είναι ε, πολύ χρήσιμο να έχουμε μία άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη δικαστική απόφαση. Ε, τώρα η απόρριψη της πρότασης είναι απόρριψη του διαλόγου. Δεν νομίζω ότι βοηθούμε αφού όλοι συμφωνούμε ότι δεν εφαρμόζεται καλά υπάρχουσα οδηγία. Ε, και η κυρία Βαν αν θέτει ε, το αίτημα του Άμλετ ε, να ζούμε ή να μη ζούμε πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε το διάλογο ή θα τον κλείσουμε. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ. Τελικά όμως έγινε ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και εγώ έχω κάποιες απόψεις να μοιραστώ μαζί σας. Ε, είχα εμπλακεί σε αυτό το θέμα ε, με μια ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών για το χρόνο ανάπαυση. Τέλος πάντων δεν θα εμπλακώ τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Ε, υπήρχε άλλη μια ερώτηση της κυρίας το προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να σχολιάσετε και αυτό που είπε ο κύριος Στιβενιούς για την απόφαση του ΔΕΚ. Να μας τα διευκρινίσετε αυτά τα θέματα. Αν θέλει, η Επιτροπή μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα δύο ζητήματα. Θέλει. Next time. Α, την επόμενη φορά, λέει η Επιτροπή. Δεν θα απαντήσει σήμερα η Επιτροπή. Λοιπόν, στις 2 Μαρτίου θα ψηφίσουμε. Θα δούμε ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά με την ε, συνολική απόρριψη της πρότασης ή αν θα υποβάλει μεμονωμένες τροπολογίες. Πάντως, λίγη συζήτηση σήμερα για αυτό το θέμα. Πάμε στα επόμενα δύο ζητήματα τώρα. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, λεπτομέρειες εφαρμογής και το παράρτημα 11 του κανονισμού. Οι συγγητές, ε, ο κύριος Κρέμες και η κυρία Λάμπερτ, πρώτη κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης ε, δεν θα συζητηθεί με τόσο πάθος όσο το προηγούμενο. Γιατί Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν τη λήξη της θητείας που είναι ο στόχος μας. Αυτό τουλάχιστον να έχουμε συζητήσει με τους σκιώδεις εισηγητής. Ένα λεπτάκι. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι τροποποιήσεις για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Νομίζω ότι τώρα πολύ περισσότεροι γνωρίζουν το θέμα εξαιτίας της οδηγίας για τη διασυνοριακή υγεία η οποία τουλάχιστον για αυτό το λόγο είναι χρήσιμη οι τροπολογίες που προτείνω για τη σύνθεση του Συμβουλίου θα δείτε ότι είναι πολύ λίγες. Ένα σημείο που προέκυψε είναι αυτό των προθεσμιών και του χρόνου που απαιτείται πολύ συχνά προκειμένου να λάβουμε απαντήσεις από κράτη-μέλη και για την επικοινωνία των κρατών μελών. Αυτό που ζητάμε είναι να προσπαθήσουν να σεβαστούν τις προθεσμίες τους στα κράτη-μέλη αλλά διαπιστώσαμε ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν δικές τους προθεσμίες. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια αναφορά στο διατακτικό του κειμένου. Προτείνω λοιπόν να έχουμε μια αιτιολογική σκέψη όπου θα αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη που έχουν δικές τους ε, προθεσμίες θα πρέπει να τις και τα υπόλοιπα να εξετάσουν την υιοθέτηση τέτοιων προθεσμιών. Επίσης υπάρχει και η ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε μετά από τέσσερα έτη να επαναξετάσουμε το σύστημα και να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και αν λειτουργεί όσο αποδοτικά και ταχύτερα θέλουμε η βάση δεδομένων για ανταλλαγή πληροφοριών. Από ό,τι μας λέει η Κομισιόνα, θα χρειαστεί το νέο σύστημα τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη οπότε θα χρειαστούμε και κάποιο χρόνο παραπάνω μέχρι να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις συνέπειές του. Και αυτό σχετίζεται και με την πρόταση του Συμβουλίου στο άρθρο 86. Ένα άλλο θέμα τώρα. Ενημέρωση των ατόμων. Αυτό θέλουμε να μπει κάπου πιο, σε ένα πιο εμφανές σημείο του κειμένου. για να γνωρίζουν τα άτομα πώς μπορούν να πληροφορηθούν. Γι' αυτό προτείνω να περάσει από το 89 παράγραφος 3 στο άρθρο 3. Υπάρχουν ε, τρεις σχετικές τροπολογίες, μία προτείνει διαγραφή, δύο άλλες προτείνουν μετατόπιση. Εγώ ενδεχομένως θα ήθελα να αλλάξει και η διατύπωση. Κάτι άλλο τώρα. Στην πρώτη ανάγνωση δεν δεχθήκαμε την άποψη του Συμβουλίου για τον τρόπο, για την περίοδο υπολογισμού γιατί θεωρήσαμε ότι είναι υπερβολικά περίπλοκη η διαδικασία υπολογισμού και για κάποια κράτη-μέλη θα χρειαζόταν υπολογισμός με βάση 365 ημέρες. Δεν είχαμε δεχτεί λοιπόν αυτόν τον τρόπο υπολογισμού, αλλά μας έδειξαν σε μένα και στους σκιώδεις εισηγητές ότι για κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Οπότε, ναι, για τα λίγα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα, αν επικεντρωθούν πλέον στις περιόδους, θα χάσουν ορισμένα άτομα κάποια συνταξιωτικά δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια του άρθρου 86 προσπαθούμε να δούμε λίγο το θέμα της ε, περίοδου υπολογισμού παρά το γεγονός ότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Αυτές είναι οι τροπολογίες που προτείνω εγώ. Βεβαίως θα προκύψουν και άλλα πράγματα μετά την εξέταση του θέματος ε, και βεβαίως θα συζητήσουμε ό,τι προκύψει και από τις απαντήσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Μετά από αυτή την εισαγωγή της κυρίας Λάμπερτ, προτείνω να ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να σχολιάσουν τη δική της νομοδότηση. Ο κύριος Κρέμερς και η κυρία Τσίμερ έχουν ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστήσω εκ νέου τον συνάδελφο τον κύριο Λάμπερτ για κύριε Λάμπερτ για το φάκελο με το οποίο ασχολείται εδώ και κάποια χρόνια Πράγματι τις τελευταίες εβδομάδες ε, ασχοληθήκαμε με κάποια άλλα ζητήματα τα οποία δεν φαίνονται στην κοινή θέση. Πράγματι οι λεπτομέρειες εφαρμογής ε, είναι πολύ σημαντικές αλλά είναι γραμμένες από την οπτική γωνία των αρχών που θα τις εφαρμόσουν και λιγότερο από τη σκοπιά των ανθρώπων που αφορούν για να μπορούν να λάβουν κάποιες πληροφορίες. Και από την πρώτη ανάγνωση λέμε πως καλό θα είναι να γνωρίζει αυτός που τον αφορά ή αυτή που τον αφορά να ξέρει σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι και προσπαθούμε να κάνουμε και μια πρόταση ανάλογη. Ένα νέο στοιχείο στην ε, κοινή θέση εδώ πέρα ε, έχει εισαχθεί από το Συμβούλιο ότι σε διάφορα σημεία δηλαδή η διατύπωση insured persons ασφαλισμένη έχει γίνει persons concerned, τα άτομα τα οποία αφορά. Ένας ορισμός ο οποίος όμως δεν υπάρχει στον κανονισμό τον, τον βασικό. Δεν υπάρχει στον κατάλογο συγκεκριμένα των ορισμών του κανονισμού αυτού. Υπάρχει μες στον κανονισμό. Η έννοια αυτή λοιπόν ασφαλισμένα άτομα, άτομα που ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να, να ξεκαθαριστεί νομίζω στην, στην ομοθεσία και θα καταλήξουμε σε μια πρόταση για να αλλάξει αυτό κάπου και να μιλάμε πράγματι για τα ενδιαφερόμενα άτομα που μπορεί να είναι είτε ο άμεσα ασφαλισμένος είτε η οικογένειά του ή η κληρονόμη. Τέλος υπάρχει ένα πρόβλημα που εκκρεμεί ακόμα και αφορά το παλαιό έντυπο ε101 το, και την αντικατάστασή του. Αυτό το οποίο κατά κανόνα πήγε, έπαιρναν οι άνθρωποι που πήγαιναν να εργαστούν για λίγο χρόνο σε άλλο κράτος μέλος για να μπορούν να βασιστούν στο ε, σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του κράτους που βρίσκονται και σε σχέση με αυτό το θέμα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να, να ξαναδούμε αλλά ε, δεν έχουμε κάποια έτσι πολύ σοβαρά ζητήματα ή αντιρρήσεις, απλά θέλουμε να δούμε κάποιες βελτιώσεις αυτή τη στιγμή στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ε, κυρία Τσίμερ και η κυρία Λίνα ακολουθούν. Äh, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λάμπερτ ε, για την ε, γνωμοδότηση της, ε, την έκθεση αυτή και να πω πως μπορούμε να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες σας γιατί στόχο έχει να φύγουμε από αυτή την ε, τυπική αντιμετώπιση του, του θέματος. Συμφωνώ εδώ και με τον συνάδελφο που μόλις μίλησε, γιατί το ζήτημα δεν είναι τελικά να κοιτάμε το ζήτημα αυτό μόνο από τη σκοπιά της διοίκησης, αλλά εντάξει, η ζωή εξελίσσεται και πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για να μπορεί ο κόσμος να κινηθεί. Οπότε πρέπει να καταλήξουμε γρήγορα σε μια κοινή θέση της ε, Επιτροπής μας. Ελπίζω να μην έχουμε εδώ πέρα μεγάλες διαφωνίες όπως το, στο προηγούμενο θέμα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Η κυρία Λίν δεν είχε ζητήσει το λόγο για άλλο θέμα, μου κάνει νόημα. Το Συμβούλιο μήπως θέλει να πάρει το λόγο. Πριν να ακούσουμε ξανά την κυρία Λάμπερτ που θα σχολιάσει παρεμβάσει των μελών της Επιτροπής. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ε, γνωρίζουμε τις συστάσεις ήδη στο Συμβούλιο Συνεδριές η σχετική αρμόδια ομάδα εργασίας ε, αυτή την εβδομάδα συζήτησε τις προτάσεις Λάμπερτ και Κρέμερς και ακούσαμε και τις πρώτες αντιδράσεις των ε, κρατών μελών. Από τις διαπραγματεύσεις λοιπόν προκύπτει πως τα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές ε, αξιολογούν θετικά τις ε, τροπολογίες αυτές ε, και το Συμβούλιο βεβαίως θέλει να συμφωνήσει με το Κοινοβουλίο στη δεύτερη ανάγνωση. Η, κατάσταση, με συγχωρείτε, τωρινή αξιολογείται θετικά, ενώ εδώ πέρα τις τροπολογίες και τροπολογίες ε, φέρνουν ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πιο κοντά σε μια κοινή λύση. Πρέπει όμως ακόμα να περιμένουμε να δούμε ποιες τροπολογίες θα υποβληθούν ακόμα γιατί έχουμε προθεσμία. Έχετε προθεσμία μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου. Οπότε θα δούμε τι θα κατατεθεί μέχρι τότε. Σε γενικέ γραμμές είμαστε θετικοί ω Συμβούλιο λοιπόν όσον αφορά τι τροπολογίε που έχουν κατατεθεί. Για την ε, Τσεχική Προεδρία τα ζητήματα αυτά τα κοινωνικά είναι προτεραιότητα και θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Και άλλο. ε... Σας ευχαριστούμε. Κυρία Λάμπερτ, έχετε σχόλια πριν περάσουμε στην έκθεση του κύριου Α, πολύ ωραία. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο παράρτημα. Το οποίο είναι αρμόδιος ο κύριος Κρέμες. Ναι κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα για την ημερήσια διάταξη. Δεν αναφέρεται εδώ πέρα προθεσμία για τις τροπολογίες αλλά βλέπω πως μου είπε η γραμματεία πως ισχύει η ίδια προθεσμία με την έκθεση της συναδέλφου Λάμπερ τώρα για το παράρτημα μπορώ να είμαι σύντομος στο παρελθόν αυτό ήταν ζήτημα δύο ξεχωριστών φακέλων που βεβαίως εντωμεταξύ μεταξύ ε, συνενώθηκαν ε, και υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την πολιτική γραμμή που επιλέχθηκε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου συγκεκριμένα για το παράρτημα 3 στην ε, θέση του Κοινοβουλίου που είναι να καταργηθεί τελείως αυτό το παράρτημα 3. Το παράρτημα 3 οδήγησε το Συμβούλιο Υπουργών σε μια νέα συζήτηση όπου πολλές βόρειες σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία τοποθετήθηκαν και δεν ε, συμφωνούσαν εξορισμού με την κατάργηση του βραχυπρόθεσμα. Οπότε από ό,τι αντιλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή θέλουμε μια ρεαλιστική τοποθέτηση οπότε μπορούμε να πούμε πως θα γίνει κάτι τέτοιο υπό όρους, ε, δηλαδή θα τονιστεί η σημασία του παραρτήματος 3 ε, και ελπίζω να μπορούν να συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα για να μην έχουμε και κάποια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο για το παράρτημα. Ο κύριος Κίκελ. Μήπως έχει να μας πει κάτι. Όχι. Πολύ ωραία. Για αυτά τα σημεία για τις εφαρμοστικές διατάξεις ε, και για το παράρτημα. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 19 Φεβρουαρίου. Και στις 30 Μαρτίου θα συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες. Και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση με το Συμβούλιο τον Απρίλιο. Λίγη συζήτηση για αυτά τα δύο σημεία. Και έχουμε ένα τελευταίο σημείο για το πρωί. Πάλι η κυρία Λάμπερτ είναι η συγγήτρια. Ε, γνωμοδότηση πρωτοβουλία για την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασία ατόμων. Κυρία Λάμπερτ, έχετε τον λόγο. Thank you, just... Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Right. The, um, ένα λεπτό να βρω το κείμενο. Η συγκεκριμένη έκθεση προέκυψε από τη διαβούλευση που έκανε πρόσφατα η Κομισιόν με αρκετές οργανώσεις από το ευρύ κοινό και από τις συστάσεις που προέκυψαν από αυτό που πήγαν στο Συμβούλιο έκανε και το Συμβούλιο δήλωση σε σχέση με αυτές τις συστάσεις. Είναι σαφές ότι ένα μέρος ε, του υπόβαθρου της στάσης τους είναι ότι αναγνωρίζουν και αυτοί ότι σε περίοδο οικονομικής ύφεσης παραμένει σημαντικό το να αποφευχθεί ο αποκλισμός ακόμη περισσότερων ανθρώπων από την αγορά εργασίας σε μακροπράθεσμη βάση. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων. Αναφέρονται τρεις περιπτώσεις στήριξη του εισοδήματος, αγορά εργασίας που δεν θα βοηθάει τον αποκλεισμό και ποιοτικές υπηρεσίες. Στην έκθεση προσπάθησα να αναφερθώ σε ορισμένες αρχές που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια των ατόμων, κάτι που τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Γι' αυτό όταν μιλάμε για στήριξη του επαρκούς ε, εισοδήματος πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ε, και το στόχο μας ε, κατά της φτώχειας εφόσον έχουμε και το έτος αντιμετώπισης της φτώχειας να έχουμε ως στόχο το να τους βοηθήσουμε να προδεύσουν. Και αυτή η συνοχιζόμενη στήριξη κατά τη μεταβατική περίοδο όπου κάποιος περνάει από τον αποκλεισμό στην προεργασιακή περίοδο που μπορεί να περιλαμβάνει κατάρτιση κτλ. Μέχρι την περίοδο της εκ νέου απασχόλησης, για όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει από όλα τα συστήματα στήριξης. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ψάχνουν για μερική απασχόληση ή κάτι αντίστοιχο και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση από τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς επίδομα ανεργίας επειδή δουλεύει μόνο Παρασκευές και Σάββατα και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τώρα όσον αφορά τα κίνητρα, που συνήθως δεν είναι κίνητρα αλλά κυρώσεις και τα οποία χρησιμοποιούν ορισμένα κράτη-μέλη, πρέπει επίσης να εξεταστούν προκειμένου να μην συγκρούονται με τις ε, συστάσεις και τους στόχους για την αντιμετώπιση φτώχειας, έτσι ώστε να μην ποινικοποιούμε την είσοδο στην αγορά εργασίας αυτών των ανθρώπων όσον αφορά τώρα την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, το τόνισαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ισχύουν βεβαίως γενικά για όλους τους εργαζόμενους, αλλά ειδικά για αυτά τα ευάλωτα άτομα πρέπει να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη και ενδεχομένως και εξατομικευμένη στήριξη γιατί υπάρχουν πολλά πολύπλοκα ζητήματα που τους αφορούν και τα οποία δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν με μια γενική και ενιαία προσέγγιση για όλους. Αυτό που τόνισε ιδιαίτερο στο Συμβούλιο είναι το θέμα της στέγασης που συχνά το υποτιμούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Όπως για παράδειγμα ακόμη και το να έχει κάποιος σταθερή μόνιμη διεύθυνση είναι πολύ σημαντικό για να επανέλθει στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε επίσης το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα σε σχέση με τα μέτρα κατά των διακρίσεων και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άτομα που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο αποκλεισμό, για παράδειγμα άτομα με ψυχολογικά προβλήματα κτλ. Ακόμη λοιπόν και τα μέτρα κατάρτισης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις πολύπλοκες ανάγκες βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη απαιτούν να υπάρχει περίοδος κατάρτισης 40 ωρών της εβδομάδα. Όταν έχουμε να κάνουμε με άτομα, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε περίοδο ανάρρωσης από σοβαρή ασθένεια και είναι πολύ δύσκολο να τους ζητηθεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση και αυτό στα πλαίσια των <coughs> προγραμμάτων Equal και του Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να υπάρξει και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενημέρωση και διάδοση των δυνατοτήτων. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Υπάρχουν ανησυχίες από διάφορες οργανώσεις με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή για το κοινωνικό ταμείο. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει όμως να περικόψουμε κάποια προγράμματα που αφορούν άλλες ανάγκες. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε μόνο αυτούς που είναι πιο εύκολο να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και να μην ασχοληθούμε με άλλες πιο δύσκολες περιπτώσεις που όμως ενδεχομένως ε, θα μπορούσαν να μας προσφέρουν πιο δημιουργικές λύσεις τελικά. Αυτά για την έκθεση. Γνωρίζω βεβαίως ότι δεν καλύπτει τα πάντα, αν και είναι περιορισμένο το πεδίο εφαρμογής. και ειδικά σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν πολλές θέσεις απασχόλησης, εμείς προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην αγορά εργασίας. Είναι αλήθεια ότι ορισμένα θέματα τα καλύπτω σε μια μισή γραμμή, όμως βασίζομαι και σε εσά ότι θα μας βοηθήσετε να διευρύνουμε αυτές τις περιπτώσεις και να επεκταθούμε. Ο κύριος ε, Φόλ στη συνέχεια η κυρία Λίνε και ακολουθούν διάφοροι άλλοι στον κατάλογο μιλητών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι βλέπω πως τα περισσότερα μέλη εδώ πέρα αποχώρησαν της Επιτροπής και έχω έτσι μια περίεργη αίσθηση. Όλο και περισσότερα έγγραφα βγάζουμε με όλο και λιγότερα αποτελέσματα. Τώρα για την έκθεση εδώ πέρα Λαμπέρ με κάθε σεβασμό προς τον συνάδελφο δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ε, γίνεται αυτή η πρόταση έχουν επαναληφθεί εκατό φορές αυτά τα πράγματα από την Κομισιόν, από το Κοινοβούλιο είχαμε ήδη τόσα έγγραφα δεν χρειάζεται πάλι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα θέλω να τονίσω πως αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη βλέπουμε μέτρα προστατευτισμού. Χιλιάδες εργαζόμενοι απολύονται και εμείς μιλάμε για έγγραφα τα οποία δεν αλλάζουν την κατάσταση. Δεν έχω κάποια τροπολογία, ελπίζω απλά να μην ε, κατατεθούν και πολλές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λίνη, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ. Μπορώ να καταλάβω αυτό το επιχείρημα σε ένα ορισμένο βαθμό, αλλά δεν θα υπερέβαλα τόσο πολύ να πω δηλαδή ότι δεν ε, κατορθώνουμε και τίποτα αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ την Τζιν που αναφέρθηκε στην μελέτη σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. Εγώ ήμουν αρμόδια στην Επιτροπή για αυτό το θέμα και εντάξει, ναι, πρόκειται για επικάλυψη ως προς πληροφορίες που δίνουμε σε μεγάλο βαθμό και ε, ε, θα νομίζω ότι θα ήταν λάθος από πλευράς μας να μην εκδώσουμε έκθεση γιατί πρέπει να τοποθετεί το Κοινοβούλιο. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, όχι επειδή ε, θεωρώ πως δεν είναι καλή η γνωμοδότηση, απλά ε, επειδή δεν είχατε πολύ χώρο, είναι δύσκολο να τα χωρέσετε όλα μέσα αυτά που θέλετε. Για την παράγραφα 6 έχω ένα σχόλιο. Ε, θέλω να αναφερόμαστε στο ελάχιστο εισόδημα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να το επιτύχουμε, δηλαδή μέσω οδηγίας, ε, δηλαδή για τον απολωτρίο το ατομικό δικαίωμα για ένα ε, κατώτατο εισόδημα σε σχέση με την ανέργεια. Στα επίπεδο κρατών μελών μάλλον πρέπει να το ορίζουμε. Ε, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η πρόταση. Αν έχουμε κάνει την αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλουμε πρόταση οδηγίε για αυτό το θέμα. Δεν το γνωρίζω. Παράγραφος 7 για τον ελάχιστο μισθό. Ε, εδώ μια αντίστοιχη φρασιολογία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όπως για το ελάχιστο εισόδημα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και πάλι να έχουμε πολιτική ελάχιστου μισθού, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ε, αυτό το θέμα της πολιτικής του κατώτατου μισθού. Ε, βέβαια, οι παράγραφοι 6 και 7 μιλάνε για δύο διακριτά ζητήματα, αλλά μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη διατύπωση. Σχετικά με την πνευματική υγεία τώρα, ε, θα ήθελα να υποβάλω κάποιες τροπολογίες για να τονίσω κάποια προβλήματα που υπάρχουν, διότι πολλοί αποκλείονται όχι μόνο από την αγορά εργασίας, ε, αλλά και από την κοινωνία γενικότερα λόγω τέτοιων ε, ψυχικών προβλημάτων. Επίσης θα υποβάλω και άλλες Τροπολογήσε για την ε, κατάχρηση συνοπνευματοδών και ε, την ε, τοξικομανία υπό ως αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού και πώς μπορούμε με βέλτιστο τρόπο να ανταλλάξουμε τις καλύτερες πρακτικές για να ενταχθούν οι τοξικομανείς και οι αλκοολικοί στην κοινωνία. Διάφορε τροπολογίε θα υποβάλω για το 14 τώρα, για την πρόσθετη στήριξη για την αγορά εργασία. Εδώ δεν καλό θα ήταν να αναφερθούμε στην οδηγία του 2000 για την απασχόληση, διότι ακόμη διάφορα κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν πλήρω και κάποια καθόλου. Οπότε. Ας το θυμίσουμε, α το υπενθυμίσουμε. Ε, ότι υπάρχει αυτή η οδηγία εφόσον μιλάμε για ενεργητική ένταξη στην αγορά εργασίας κυρίως με αποδέκτες τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν την οδηγία και θα κινηθούν διαδικασίες επί παραβάση εναντίον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τσίμερ και μετά η κυρία Παναγιωτοπούλου Κασιώτου. Mm. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τζιν Λάμπερτ για την έκθεση αυτή και για το ότι υπέβαλε μια έκθεση η οποία κατά την άποψή μου είναι πολύ ωραία και την υποστηρίζω σε βασικές κατευθύνσεις. Για δύο πράγματα θα ήθελα να πω κάποια λόγια. Πρώτα απ' όλα Έχουν ε, γίνει εδώ πέρα κάποιες τροπολογίες ε, που είναι προσθήκες και μπορούν να κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο αυστηρά ή τα κάνουν πιο συγκεκριμένα και κυρίως με στόχο να έχουμε πιο συγκεκριμένους στόχους για να ξέρουμε και τι, τι θέλουμε εδώ πέρα. Να έχουμε δηλαδή συγκεκριμένους στόχους για να ξέρουμε μετά και που, που βαδίζουμε όσον αφορά την καταπολέμηση της στόχιας από τα κράτη-μέλη για να μην λέμε τα ίδια. Και το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι πως ευχαριστώ την Τζιν Λάμπερτ για την διατύπωση που έχει στο άρθρο 10 και 18 γιατί εδώ κατά την άποψή μου ξεκαθαρίζει ε, το ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα ειδικά γιατί οι άνθρωποι δεν καταντάσσονται πάντα στις κατηγορίες που, και στις ετικέτες που εμείς θέλουμε να τους βάλουμε. Εγώ έχω μία εμπειρία πως υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες ανθρώπων, τους οποίους εμείς ε, προσπαθούμε, η κοινωνία προσπαθεί να δημιουργήσει ε, συνθήκες ένταξης, αλλά μπορεί να αποτύχει αυτή η προσπάθεια. Και δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως μπορεί πάντα να υπάρξει αυτή η ενσωμάτωση. και είναι προσανατολισμένη και η πολιτική απασχόληση και η κοινωνική πολιτική να χρηματοδοτεί έργα που στοχεύουν προς, αυτή την ένταξη στη διαδικασία της εργασίας. Και η κυρία Λάμπερτ γράφει ε, προσεγγίσεις προς την επανένταξη διατρέχουν τον κίνδυνο να μην χρηματοδοτηθούν. Μπορεί σε κάποια κρατημέλη, αλλά αλλού ίσως να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση ή να είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα ε, έργα αυτά για να επιτύχουν τίποτα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί καμιά φορά απλά για έξι μήνες ε, τους βγάζουμε από την δινή τους κατάσταση και μετά ξαναπέφτουν εκεί που ήταν πριν και δεν υπάρχει καμία δομή και τίποτα άλλο. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το ε, τονίσουμε και να πούμε πως οπωσδήποτε δεν πρόκειται ε, ε, οπωσδήποτε για ανθρώπους ε, μόνο με αναπηρία. Δεν μιλάμε για κάποιες ανθρώπους που υφίστανται διακρίσεις. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάποια εμπόδια τα οποία είναι δύσκολο να τα υπέρβουν. δηλαδή μακροχρόνια άνεργοι, άνθρωποι που δεν έχουν κοινωνικές ικανότητες, που έχουν ψυχολογικά προβλήματα που μπορούμε, πρέπει να βρούμε τελείως διαφορετικές λύσεις και να δικτυωθούν περισσότερο αυτά τα έργα για να έχουμε μια κοινωνική, παιδαγωγική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη και να, μπορέσουμε, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν στην κοινωνία ακόμη και αν δεν έχουν τελικά τη δυνατότητα να εργαστούν και να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Αυτά ε, είναι η ουσία των τροπολογιών που έχω βάλει. Ευχαριστούμε. Πολύ γρήγορα ε, θέλω να ε, πω ότι δεν έχουν, έχει δίκιο ο συνάδελφος που αποχώρησε και από την αίθουσα να θεωρεί περιττές τις συζητήσεις ή περιττή την ενασχόληση με τέτοια θέματα έστω και αν επαναλαμβανόμεθα ε, είναι απολύτως απαραίτητο και μέσα στα καθήκοντά μας να συνεχίζουμε να προτείνουμε λύσεις Βέβαια οι λύσεις αυτές δεν πρέπει να είναι λύσεις κλισέ. Ε, φαίνεται πολλές φορές και από τις τροπολογίες μας και είναι λυπηρό ότι έχουμε κάποιες σταθερές ιδέες. Είναι ε, κίνδυνος να θεωρηθεί ότι έχουμε και έμονες ιδέες που τις επαναλαμβάνουμε στις ε, τροπολογίες μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ευέλικτες λύσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους ότι ο άνθρωπος αλλάζει και ότι μπορεί να πέσει από τη μία κατάσταση στην άλλη και να έχουμε έτοιμες υποδομές που θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αντιμετωπίζουν αυτές τις αλλαγές ε, που έρχονται και με την ηλικία και με την αλλαγή ε, των οικονομικών ε, συνθήκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πράγματι περίπλοκο το ζήτημα και δεν πρέπει να κατηγοριοποιούμε αλλά να δημιουργούμε υποδομές έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίζουμε και αυτούς που σταθερά αποκλείονται και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι μερικοί σταθερά αποκλείονται από την αγορά εργασίας αλλά να δημιουργούμε και τη δυνατότητα για όσους μπορούν να μεταπηδήσουν στην κατάσταση του ενεργού εργαζόμενου να μπορούν να το κάνουν όποτε ε, αυτό είναι δυνατόν. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να ε, ε, υποθέτουμε είναι ότι μπορεί να δοθούν λύσεις μέσω οδηγιών. Οδηγιών για το ελάχιστο εισόδημα ή οδηγιών για το κατώτατο μισθό. Αυτά δεν γίνονται με οδηγίες, γίνονται μόνο με την σύνθεση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης γιατί για την αξιοπρεπή διαβίωση δεν φτάνει μόνο ένα κατώτατο εισόδημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλον δεν έχουμε στον κατάλογο μιλητών, οπότε... Ο, ο κύριος Καλαντρίνο από πλευράς Επιτροπής θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη της Επιτροπής. Ε, για την σημερινή μας συζήτηση καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, ε, γνωμοδότηση αυτή Εξ αρχής ο κεντρικός ρόλος και η σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναγνωρίστηκε από πλευράς μας για αυτήν την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας. Ήδη στην ανακοίνωση 620 του 2007 όπου δρομολογήθηκε το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων για την πρωτοβουλία για την ενεργητική ένταξη. Η Επιτροπή Εισηγήθηκε την έγκριση κοινών ε, αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα της ένταξης και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί και το έρισμα για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και για ε, ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Κοινέ αρχές λοιπόν και κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, στις 3 Οκτωβρίου του 2008 στην σχετική ανακοίνωση το Συμβούλιο το Δεκέμβριο ενέκρινε τα, τα συμπεράσματά του συγγνώμη, και καλωσορίζουμε αυτήν την γνωμοδότηση από πλευράς ε, του Κοινοβουλίου, από το τρίτο θεσμικό όργανο της Ένωσης, δηλαδή για αυτό το τομέα. Θα σας θα κάνω μία διευκρίνηση μόνο για τον ορισμό και τη λογική που διέπει αυτή την πρωτοβουλία και να τονίσω ε, τρία στοιχεία που μας υπέδειξε η συγγήτρια και να μιλήσω για τα μελλοντικά βήματα. Λοιπόν, η πρωτοβουλία για την ενεργητική ένταξη δεν είναι μια απλή πρωτοβουλία για την ένταξη των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Εάν δούμε την πρώτη παράγραφο των συστάσεων του Οκτώβρη, βλέπουμε το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας και λέει εκεί ότι οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης πρέπει να διευκολύνουν την ένταξη σε βιώσιμη ποιοτική απασχόληση για όσους μπορούν να εργαστούν και ε, παροχή παρκών πόρων για να ζουν όλοι αξιοπρεπώς ε, σε συνδυασμό με ε, την κοινωνική συμμετοχή όλων όσων δεν μπορούν να εργαστούν. Δηλαδή όλοι όσοι αποκλείονται από την αγορά εργασίας είναι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας και υπενθυμίζω ότι η νομική βάση για τις συστάσεις ε, είναι το άρθρο 137H ε, της ε, συνθήκης ένταξη των ανθρώπων που έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας είναι στρατηγική για όλους, δηλαδή που, έχουν, που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι οι δύο δρόμοι υπάρχουν ε, για την ένταξη. Πρώτον, πρέπει να προάγουμε την ένταξη σε ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση για όσους μπορούν να εργαστούν για να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια, αλλά να γνωρίζει η ανακοίνωση επίσης ότι αυτό δεν είναι βιώσιμη αλλακτική λύση για όλους και άρα πρέπει να παράσχουμε πρόσβαση σε επαρκή στήριξη εισοδήματο για όλους και ευκαιρία για κοινωνική συμμετοχή, συμμετοχή στα κοινά. Ε, μάλλον κοινωνική συμμετοχή, κάτι που η Επιτροπή των Περιφερειών τόνισε πάρα πολύ στη σχετική γνωμοδότησή της. Και ακόμη και όσοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, θα πρέπει τουλάχιστον μπορούν να συμμετάσχουν ε, στην ε, κοινωνία μέσω εθελοντικής εργασίας να έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες του τομέα της υγείας, ε, δηλαδή αποκατάσταση, κατάρτιση για όλους, ε, δηλαδή ούτως ώστε όλοι να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία στην οποία ζουν. Σε σχέση με την πρώτη παρέμβαση που ακούσαμε θα προσθέσω το εξής. Υποβάλαμε αυτή την πρόταση διότι αυτή αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη νομική πράξη που υποβάλλει η Επιτροπή ε, για το θέμα της κοινωνικής ένταξης. Μετά τη συμπερίληψη στη συνθήκη του Άμστερνταμ το 97 των κοινωνικών διατάξεων, που εγκρίθηκαν βέβαια το 99, αυτό είναι λοιπόν το πρώτο νομοθέτημα στον τομέα της κοινωνικής ένταξης. Ε, δηλαδή πρώτη ε, απτή χρήση, εφαρμογή των κοινωνικών διατάξεων. Οπότε ε, μπορεί να ισχυριστεί το Κοινοβούλιο ότι είναι λίγο ε, ισχνό το, το, το νομικό αυτό εργαλείο, αλλά παρόλα αυτά συνιστά ε, σημαντικό βήμα προόδου και υπάρχει μια ιεράρχηση. Έχουμε εγκρίνει τις συστάσεις και ε, που ακολούθησαν την αρχική ανακοίνωση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της κοινωνικής ένταξης ε, στις μέρες μας γιατί όλο ένα και περισσότερο δυσκολεύονται να συμμετάσχουν όλοι στην αγορά εργασίας και να έχουν ένα επαρκές εισόδημα. Οπότε Θα τονίσουμε και πάλι αυτή την πτυχή και σε συνδυασμό φυσικά με την ε, οικονομική κρίση που βιώνουμε. Τώρα, ε, για την ουσία τρει παρατηρήσεις. Η αιρεσιμότητα. Ε, συμφωνούμε με την εισηγήτρια, είναι πολύ λεπτό το θέμα και την ανακοίνωση την προετοιμάσαμε από κοινού με ε, τα κράτη-μέλη έγιναν διαβουλεύσεις μέσα από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα. Απλά ήθελα να τονίσω πως Πρέπει να υπάρχει μια αιρεσιμότητα ούτως ώστε να μην απαγιδευτούν στις παροχές ε, ε, όλοι. Δηλαδή μέσα σε αυτή την ανακοίνωση δεν αποσκοπούμε σε, στο να έχει κάποιος ε, οπωσδήποτε πάση θυσία μια θέση απασχόλησης. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ενεργή διαθεσιμότητα είτε για απασχόληση είτε για επαγγελματική κατάρτιση για όλους όσους δεν μπορούν να εργαστούν. Δηλαδή Υπάρχουν δύο εναλλακτικέ. Αν μπορεί κάποιο να εργαστεί, να εργαστεί, αλλιώ να ε, ε, υπάρξει επαγγελματική κατάρτιση και συνδυάζεται με άλλα μέτρα κοινωνική ένταξη. Ε, δηλαδή, υπάρχει αυτό ο δυνητικό χαρακτήρα που σα περιέγραψα. Τώρα, ε, είναι ένα θέμα που απασχόλησε πολύ τη Γαλλική Προεδρία, δηλαδή η υποστήριξη μέσα στην αγορα εργασία, εργασίας, in-work support. Ε, έχουμε το Γεβενίντο Solidarity Active, το σχετικό σύστημα στην ε, Γαλλία. Ε, εισόδημα αλληλεγγύης όπως ονομάζεται, δηλαδή υπάρχει υποστήριξη και εκτός και εντός αγοράς εργασίας και έχουμε τις τέσσερις βασικές αρχές σε σχέση με την ενεργητική ένταξη στην αγορά εργασίας ε, πρέπει να προωθούνται οι ποιοτικέ θέσει απασχόλησης αλλά και να υπάρχει καταβολή των επιδομάτων ε, για να, μην, για να καταβολούμε τη φτώχεια μέσα στην αγορά εργασίας. Ε, τρίτον, το θέμα της στέγασης, ε, ρηξικέλευθο στοιχείο, αν μπορώ να το θέσω έτσι, σε σχέση με τη σύσταση του 92, Το το Συμβούλιο δεν ε, είχε καλύψει το θέμα της στέγας και των σχετικών επιδομάτων κοινωνικές αιστείες και τα, εργατικές κτλ. Τώρα όμως αυτό το θέμα εντάχθηκε στον στον τρίτο πυλώνα ε, και ε, υπάρχει η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας όπου τα κράτη-μέλη έχουν ε, θεωρήσει ότι για την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού το 2009 θα είναι η χρονιά του της ενεργητικής κοινωνικής ένταξης και κυρίως το θέμα της ε, στέγασης ε, και σας λέω θα υπάρξει συνεργασία του Κοινοβουλίου με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ε, ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για αυτό το θέμα. Τώρα για τα μελλοντικά βήματα, γιατί αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που τονίζονται μέσα στην γνωμοδότηση. Ο στόχος ε, της ε, σύστασης ήταν εν μέρη να επικαιροποιηθούν οι συστάσεις του 92 για την ε, κοινωνική αρρωγή, να τα, εγγράψουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να ενσωματώσουν και άλλους δύο ε, πυλώνες που θα μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση αυτών των μειονεκτημάτων. Ποια είναι η διαφορά με το 92, τώρα έχουμε σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης ε, της εφαρμογής ε, των ε, συστάσεων, δηλαδή την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Την ερχόμενη εβδομάδα η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα το συζητήσει το θέμα, τα μελλοντικά βήματα δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Και το Μάρτιο κατά πάσα πιθανότητα η ομάδα εργασίας ad hoc της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την κοινωνική ένταξη θα συνεδριάσει και πάλι για να συζητήσει τα μελλοντικά βήματα και ξανά στις 24 Απριλίου στην πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα ξανασυζητηθεί το θέμα. Τώρα, η υποομάδα κοινωνικής ένταξης της Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας σε διάφορες συνεδριάσεις έχει ήδη εκπονήσει ένα πρόγραμμα εργασίας για να συζητηθούν οι δείκτες του το τομέα αυτού, παραδείγματος χάρη πρόσβαση σε επαρκή στέγαση, ε, μετάβαση προς την αγορά εργασίας, ε, πρόσβαση υγειονομικές υπηρεσίες, ε, συστήματα κατοχύρωσης ελαχίστου εισοδήματος, ε, και οι υπηρεσίε ε, τη επιτροπή θα παρακολουθούν ε, συστηματικά και την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Έχουμε και τον εξάρτητο δίκτυο των εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική ένταξη που θα συντάξει επίση έκθεση για τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματο. και έχουμε και διάφορε άλλε πρωτοβουλίε που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Progress και κυρίω θα ήθελα να τονίσω το δίκτυο των παρατηρητηρίων των τοπικών αρχών για την κοινωνική ένταξη που τώρα θα ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα αρχίσει να τρέχει την 1η Μαρτίου 2009 υπό το συντονισμό των Eurocities ε, και η πρώτη πιλωτική φάση θα διαρκέσει 1,5 χρόνο και θα υπάρξουν πέντε. Στο, σε διάφορες ε, πόλεις όπως το Southampton, η Μπολόνια θα, θα δημιουργηθούν εκεί παρατηρητήρια τοπικών αρχών για την κοινωνική ένταξη ε, σε τοπικό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι θα, συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν ε, σε αυτή την πρωτοβουλία ε, για την εφαρμογή των δράσεων για την κοινωνική ένταξη. Θα σταματήσω εδώ, αλλά έχουμε διάφορα προγράμματα, αξιολόγηση από ομότιμους, peer review και άλλες πρωτοβουλίες που τρέχουν ήδη. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει από πλευρά του ε, την ε, επαρκή παρακολούθηση αυτών των τεσσάρων αρχών που σα περιέγραψα στην αρχή της παρέμβασής μου. Ευχαριστώ. Θα κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Στην συνεδρίαση των συντονιστών συμφωνήσαμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία γνωμοδότηση πρωτοβουλίας. γιατί έχουμε συζητήσει επανειλημμένα αυτά τα ζητήματα. Απλά αυτό είναι το ισχυρότερο ή μάλλον το μοναδικό ε, νομικό εργαλείο που υπάρχει στον τομέα αυτό. Και ε, γι' αυτό θέλαμε και εμείς να εκφέρουμε άποψη αυτή τη φορά συχνά επαναλαμβάνουμε τις θέσεις που έχουμε εκφράσει στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορούσαμε παρά να το κάνουμε εκ νέου, διότι ε, έχουμε τώρα την ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτό το εργαλείο που σας έλεγα, αυτή την νομική πράξη, άνευ προηγουμένου στον τομέα αυτό, η κυρία Λάμπερτ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και την ενημέρωση που πράγματι μας βοήθησε πάρα πολύ και ελπίζω ο κύριος Φάρμπερ να θεωρήσει πως η συμπερίληψη της πράγας στα παρατηρητήρια είναι συγκεκριμένο μέτρο. Εντάξει, ε, καταλαβαίνω αυτό που λέει, αλλά υπάρχει και ένα όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη. Γιατί πολλά από αυτά σχετίζεται και με το πώς χρησιμοποιούμε το Ταμείο Συνοχής ε, και τα λοιπά ταμεία και τα οικονομικά μέσα που έχουμε και τα μέσα πολιτικής. Δηλαδή το πλαίσιο έτσι ακούγεται πολύ ωραίο αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι. Ε, όσον αφορά κάποια από τα ζητήματα τα οποία ετέθησαμε το θέμα για το βασικό μισθό. Βλέποντας και κάνοντας. Θα, δηλαδή θα δούμε πώς θα κινηθούμε, αλλά είναι σαφές πως απασχολεί πάρα πολύ τα, τα κράτη-μέλη. Ε, τι υποτίθεται ότι πρέπει να καλύπτει το ελάχιστο εισόδημα για να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι συμπεριλαμβάνονται στην κοινωνία και δεν είναι στο περιθώριο. Ε, αυτό νομίζω θα είναι πρόβλημα που θα οξυνθεί τους ερχόμενους μήνες, ίσως και χρόνια. Οπωσδήποτε καλοδεχούμενες τροπολογίες μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα, αλκοολισμό, ναρκωτικά και συγκεκριμένους στόχους. για να γίνουν τα πράγματα και πιο συγκεκριμένα. Και προφανώς και η οδηγία της απασχόλησης έχει σχέση και με τον αποκλεισμό από την ε, αγορά εργασίας αλλά και με την συμπερίληψη την ε, κοινωνική, τις γενικές αρχές τουλάχιστον. Οπότε αναμένω τις τροπολογίες και φαντάζομαι θα μας υπενθυμίσει ο πρόεδρος ποια είναι η προθεσμία. Και ίσως θα μπορούσαμε να γεμίσουμε και κάποια κενά που πράγματι συνειδητοποίησα μετά από αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν ότι έχει η έκθεση. Οπότε σας ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι να δω εδώ τι σημειώσεις μου. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 16 Φεβρουαρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι. πέρας της συζήτηση και για αυτό το θέμα. Στις 2 Μαρτίου θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και αναμένεται να ε, ψηφίσουμε στις 31 Μαρτίου στην Επιτροπή μας ε, γιατί έχουμε και την ε, Ολομέλεια του Μαΐου όπου θα γίνει ψηφοφορία για αυτή την νομοδότηση. Λοιπόν, πέρα των εργασιών για το πρωί, επιστρέφουμε στις 3. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε το απόγευμα. Καλή όρεξη.